So, hallo, guten Tag. Selbst wenn noch nicht alle da sind, möchte ich gerne beginnen. Ich begrüße die Kollegen. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει όλοι, πάντως θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θέλω να καλωσορίσω τους συναδέλφους μου και τους εμπειρογνώμονες για το δεύτερο μέρος της απόψινής συνεδρίασης. Ας ξεκινήσουμε όμως ε, να καλωσορίσω την κυρία Ξελντεβό, τον κύριο Ντόχερτη, Είχε ζητηθεί από την Επιτροπή μας μια μελέτη για την εξέλιξη του διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Θα ακούσουμε σήμερα τη σχετική παρουσίαση. Θα γίνει δηλαδή μια επισκόπηση της Κομισιόν, της, της ε, ανακοίνωσής της του Απριλίου 2009 για τον εξυγχρονισμό των σχέσεων ε, πανεπιστημίων ε, επιχειρήσεων. Το Φόρουμ Διαλόγου Έχετε αναλύσει λοιπόν, ελπίζω, το διάλογο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα προσπαθήσετε να προσδιορίσετε την περαιτέρω συμβολή που θα μπορούσαμε να έχουμε σε έναν επικοδομητικό διάλογο. Η κυρία λοιπόν Ντεβό θα σας κάνει μια παρουσίαση με PowerPoint και νομίζω ότι έχετε λάβει όλοι το έγγραφο, τη σχετική μελέτη. Πριν όμως διαβάσετε το έγγραφο, κοιτάξτε και ακούστε, γιατί είναι έτσι και πιο ζωντανό. Καλό είναι λοιπόν να ακούσουμε την ε, κυρία Ντεβό 10 λεπτά το πολύ. Um, uh, Madam Chairman, Uh, Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Να σας μιλήσω για το διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και να σας παρουσιάσω τα πορίσματα της μελέτης μας. Την έρευνα αυτή εκπώνησε η Deloitte, αλλά δεν θα ήταν εφικτό κάτι τέτοιο χωρίς την συμμετοχή πολλών άλλων φορέων στο διάλογό μας, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ξεκινήσω την, την παρουσίασή μου με το ιστορικό του διαλόγου αυτού για να σας εξηγήσω γιατί η ανώτατη εκπαίδευση και τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μαζί με τις επιχειρήσεις πρέπει να συνεργάζονται. Γιατί λοιπόν ένας τέτοιο διάλογος επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Επειδή ο παγκόσμιος ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονο σε όλου του τομείς, ιδίω καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο ο κόσμο πλήττονται από την οικονομική ύφεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ενεργή και να, να προβλέψει τις ε, μελλοντικές προκλήσεις. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες των επαγγελματιών θα ε, συνάδουν με τις ανάγκες της ε, σύγχρονης αγοράς. Έτσι λοιπόν, επιχειρηματικό κόσμο και τα πανεπιστήμια πρέπει να συνεργάζονται. Αυτό είναι ο στόχος του διαλόγου μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Δεν είναι όμως εύκολο να υπάρξει συνεργασία λόγω της ποικιλία και του οικονομικού και του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού σκηνικού και τοπίου στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα η ποικιλία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πολύ συχνά έχουμε πανεπιστήμια αλλά υπάρχουν και πολυτεχνικές σχολές και επαγγελματικά Ινστιτούτα, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επίσης υπάρχει διαφορά μεταξύ στη δράση και το μέγεθο των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο διάλογο αυτό, καθώς πολλές φορές ε, είναι κινητήριο δύναμη των τοπικών, των τοπικών οικονομιών. Επίσης, ο διάλογος μας υποχρεώνει να ασχοληθούμε και με ε, τομείς όπως η διδασκαλία, Τώρα, στην ανακοίνωση του 2006 ανακοινώθηκαν ε, οι πρώτοι στόχοι του διαλόγου αυτού που ετοπίζει τομεί δράσεως για την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ατζέντα της αύξησης ε, της απασχόλησης. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού τομέα και ε, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η πρώτη φάση αυτού του διαλόγου έλαβε χώρα το το Φεβράριο του 2008 και η δεύτερη το Φεβράριο του 2009. Η ανακοίνωση του 2009 παρουσίασε τα βασικά επιτεύγματα του διαλόγου αυτού στα αρμόδια φόρα και πρότεινε μελλοντικέ δράσει ε, μέσω των συστάσεων των ε, φόρα αυτών. Η ανακοίνωση έχει διευθωθεί κατά τέτοιο τρόπο που ε, ουσιαστικά στηρίχθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους βασικούς φορούς. Υπήρξε ανάγκη για κεντρική διαχείριση του συστήματος, ώστε η όλη διαδικασία να διεξαχθεί ομαλά. Όμως ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να αποδώσει εάν τον ε, στηρίζει μόνο η Επιτροπή. Και τα κράτη-μέλη και η περισσότερη συμμετοχή των ε, ενδιαφερομένων εταίρων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα του διαλόγου. Πιστεύουμε ότι ιδιαίτερος πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κατάλληλο επίπεδο για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του διαλόγου. Λόγου χάρη πάρει. Δραστηριότητες όπως ο συντονισμός, οι ανακοινώσεις, η προώθηση, ο έλεγχος της προόδου και η υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο θα πρέπει να είναι βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει των συμβολών που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Η διαδικτύωση, η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η οργάνωση των εκδηλώσεων προώθησης και διαφήμισης θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι παράγοντε εμπλέκονται σε όλα τα επίπεδα στον κατάλληλο βαθμό, είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η προστεθέμενη αξία αυτού του διαλόγου. Οι συζητήσει στα φόρα διοργανώθηκαν βάσει έξι προτεραιοτήτων, έξι κυρίαρχων αξώνων. Πρώτα απ' όλα, στοχεύσαμε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τι επιχειρήσει και του πολίτε ακόμη και αν η παγκόσμια οικονομία μπορεί να ωφεληθεί από την περισσότερη και την καλύτερη έρευνα, οι επιχειρήσει είναι κύριοι δικαιούχοι τη ε, εύρυθμη συνεργασία όταν μιλάμε για την μεταφορά τη γνώση. Οι πολίτε και ιδίω κατά την έβρεση εργασίας θα ωφεληθούν από την πρόσβαση στα ε, CV που μπορεί να παρέχονται online στο διαδίκτυο και να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά μαζί με την ε, διαβίου εκπαίδευση. Επίση, όσοι ασχολούνται με τι επιχειρήσει ε, θα μπορούν ε, να γνωρίζουν τι επιχειρησιακέ δεξιότητε του καθενό πριν εκπονήσουν τι μελέτε του. Η συνεργασία με τι επιχειρήσει θα βοηθήσει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επιτύχουν καλύτερα του στόχου του. Ιδίω ο τομέα προτεραιότητα τη κυβέρνηση των πανεπιστημίων θέλει να δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον για να γίνει η συνεργασία αυτή πιο αποτελεσματική. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσει και οι πολίτε ε, είναι, αντικείμενο, είναι στόχο πολλών πρωτοβουλειών. Πρωτοβουλίε που αναφέρονται στη διαφάνεια που βλέπετε εδώ, τι οποίε ε, διεξάγουν οι Γενικέ Διευθύνσει για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση, για την Περιφερειακή Πολιτική, για την Έρευνα, καθώ και τι επιχειρήσει και τη βιομηχανία άλλες γενικές διευθύνσεις όπως του περιβάλλοντος επίσης συμμετέχουν σε ανάλογες δραστηριότητε. Η οριζόντια διάσταση του θέματος αυτού ε, είναι ορατή και εκτός Επιτροπής. Όπως αυτό το σώμα η παρουσίαση αυτή οργανώθηκε από την Επιτροπή σας ε, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης αλλά και οι Επιτροπές ε, Βιομηχανίας και Έρευνας υπέβαλαν εκθέσει για την ανακοίνωση τη Επιτροπή το 2009. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ευρύτατο ενδιαφέρον για το όλο θέμα. Η βασική Οι βασικοί στόχοι του διαλόγου, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και οι πολίτες είναι, αυτοί, είναι οι πρώτοι στόχοι που σας ανέφερα, αλλά ο διάλογος δεν αφορά μόνο αυτούς. Υπάρχουν και οι διαμεσολαβητές. Εδώ έχουμε παριθμίσει έναν κατάλογο συμμετεχόντων στο διάλογο, τους οποίους ε, ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της μελέτης μας για να έχουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Ποιο είναι ο ρόλο τώρα των διαμεσολαβητών αυτών των φορέων και παραγόντων. Πρέπει να εμπλέκονται ω ένα σημείο διαπαφή μεταξύ των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων. Ιδίω θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διάδοση των καλών πρακτικών, τον εντοπισμό των νέων παραδειγμάτων καλών πρακτικών που πρέπει να ακολουθούνται και την στήριξη των οργανώσεων που θέλουν να ε, ξεκινήσουν τη συνεργασία. Οι φορείς αυτοί επίσης θα πρέπει να διαματίσουν ρόλο στο να έρθουν σε επαφή με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο. Για να ολοκληρώσω αυτή την παρουσίαση, θα συνοψίσω τις βασικές συστάσεις της μελέτης μας, Επικεντρωνόμενη στην στρατηγική και επιχειρησιακή διάσταση του διαλόγου. Στο στρατηγικό επίπεδο είδαμε ότι ο διάλογος δεν περιορίζεται σε δραστηριότητε που φέρουν εις πέρας η αρμόδια γενική διεύθυνση και η επιτροπή σας στο Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις του διαλόγου και να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά ε, γνωστοποιούνται στο υψηλότατο πολιτικό επίπεδο. Επίσης, κλειδί για την επιτυχία του διαλόγου είναι πρώτον η έντονη συμμετοχή όλων των φορέων, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Έπειτα, το να είμαστε ανοιχτοί στα παραδείγματα καλών πρακτικών που έρχονται εκτό Ευρώπη, όπω από τι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει την προσπάθειά της να ενισχύσει το διάλογο και να ενθαρρύνει ακόμα περισσότερους να συμμετέχουν σε αυτόν. Ευχαριστώ. Ε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διαγκό. Δεβό. Μας δείξατε πώς θα έπρεπε να είναι ο διάλογος, με ποιον θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το διάλογο και τι δυνατότητα έχει η έννηση σε σχέση με τα διάφορα προγράμματα που αναφέρατε, το lifelong learning, το διαβίου εκμάθηση κλπ. κλπ. Για μας το σημαντικό είναι να ξέρουμε και ποια είναι τα δεδομένα, αλλά να δούμε και το περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για αυτό το πλαίσιο που μας θέσατε και θα ήθελα αν μπορούσε η Κομισιόν σύντομα η κυρία Μπενάλντο Δικοέρος αν είναι παρούσα να πάρει το λόγο την παρακαλώ και παρακαλώ να είστε σύντομοι να σχολιάσετε αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά και συμφωνούμε απόλυτα ε, με τα συμπεράσματα. Ε, ήδη συμφωνήσαμε και με τα πρώτα λόγια της εισηγήτριας ε, να υπάρχει στήριξη δηλαδή. Αυτό το τονίσαμε και εμείς στην ανακοίνωσή μας. Πρόθεση του διαλόγου, συμμετοχή του διαλόγου αυτό είναι πολύ σημαντικό και ε, θα σας πω και πώς μπορούμε να το κάνουμε απαντώντας στην έκθεση του κ. Σμιθ. Και όπως γνωρίζετε, ε, δραστηριοποιούμαστε ιδιαίτερα σε μια σειρά νέων ε, θεμάτων και νέων οδών που είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με αυτή την έκθεση, με αυτή τη μελέτη. Ίσως δεν θα έπρεπε να κάνουμε προτάσεις, αλλά να αναγνώσουμε σε τρεις στήλες την μελέτη που την παρουσίαση μόλις ακούσαμε και που είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. Έχουμε και τη δεύτερη μελέτη των καλών πρακτικών και την μελέτη την τρίτη του ETF για τις ε, Χώρε ε, τη πολιτικής γειτονία. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες, αυτές είναι οι τρεις μελέτες που νομίζω θα μας επιτρέψουν μια συγκριτική μελέτη και θα εμπλουτίσουν πολύ την ε, ανάλυση μας. Θέλω να συγχαρώ την συγγήτρια για το ποιοτικό τη έργο. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Μπενάλο Ντεκουέρος, δεν ήταν η συγγήτριά μας. Δεν είναι η συγγήτριά μας. Μετά θα μιλήσει και ο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε σε καλό δρόμο. Να συζητήσουμε σε βάθος τα θέματα αυτά. Και δεν είναι θέμα μόνο της Επιτροπής Πολιτισμού. Αφορά και την Επιτροπή Ήτρα, την Επιτροπή Ενέργειας, Έχουμε τον κύριο Πάρ Σμιτ, που είναι της Επιτροπής μας, εισηγητής και την κυρία Ρέρα Μαντουρέρ από την Επιτροπή Ενέργειας. Θα τους ακούσουμε και τους δύο. Θα μας μιλήσετε για το σχέδιο της έκθεσή σα σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Και μετά θα κάνουμε μια σύντομη συζήτηση και θα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε και σε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 Θα μιλήσω ουγγρικά. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω στην ακρόαση αυτή και να κάνω μια αναφορά στο κείμενο. Η εκπαίδευση στην Ευρώπη αλλάζει και στόχος είναι η προσαρμογή των πανεπιστημίων στο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερες ανάγκες των πολιτών ε, και των όλων της Ευρώπης. Η στατική της Λισαβόνας βέβαια ε, ολοκληρώνεται και ίσως τα αποτελέσματά της να μην μας ε, ικανοποιούν ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσουμε το πρόγραμμα 2020 να το επικεντρώσουμε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, διότι χωρίς ε, αυτές τις πτυχές δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία απασχόληση. Οι στόχοι της διαδικασίας της Μπολόνιας ξεκολουθούν να είναι έγκυροι μεταξύ αυτών δεν μπορώ να του επισημάνω όλου του στόχου, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ε, τη οικονομία και τη ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να γίνουν κοινέ προσπάθειε, οι οποίε θα διέπονται από την αρχή ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι ανοιχτά και να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό ήταν η αλήθεια από την εποχή του Μεσαίωνα. Δηλαδή τα πανεπιστήμια ε, είχαν σχέση μεταξύ τους και θα πρέπει τα πανεπιστήμια να, είναι, να έχουν ηγετική στάση και σήμερα στην Ευρώπη. Η Κομισιόν ε, πέρυσι έκανε δύο πολύ σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή προσπαθώντας να συμβιβάσει κάποιες φορές αντικρουόμενες παραδόσεις, ε, συμφέροντα, πηγές και πολιτικές από τα διάφορα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και πέρυσι εκδώσαμε αρκετές μελέτες, διοργανώσαμε και ακροάσεις σε σχέση με την ανώτερη εκπαίδευση, μία εκ των οποίων είναι και η έκθεση που έχετε ενώπιόν σα, Ένα στάδιο στην όλη διαδικασία για την σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πιστεύω ότι το θέμα είναι επίκαιρο, διότι βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δώσουμε νέα πνοή οικονομίες και να στην οικονομία και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ καλά πτυχία τα οποία δεν μπορούν να βρουν καλές θέσεις ε, αντάξει των προσόντων τους και έχουμε ταυτόχρονα όμως και πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας. Η Επίτροπος ε, στην διάρκεια της δικής της ακρόασης είπε ότι το 50% και σε κάποια κράτη-μέλη το 80% των αποφύτων δεν βρίσκουν τα πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών του σπουδών μια θέση εργασίας και αυτό σίγουρα ε, δημιουργεί σε αυτούς σημαντικά προβλήματα αλλά και μειώνει σημαντικά τις δυνατότητες αυτών των να στην αγορά, να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Ίσως ένα ζήτημα είναι η ποιότητα των τίτλων σπουδών. Μήπως υπάρχει πρόβλημα με τη διδακτέλη των πανεπιστημίων, μήπως δεν καλύπτει τις ε, απαιτήσει της αγοράς ή μήπως ο ιδιωτικό τομέα έχει πολύ ψηλέ ε, προσδοκίες και απαιτήσει από τους αποφύτου. Οι επιχειρήσει συνήθως ε, μπορούν να συνεργαστούν με την εκπαίδευση εκεί που υπάρχει άμεσο όφελος και κέρδος, έρευνα και ανάπτυξη για παράδειγμα που μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις ή ε, κάτι άλλο. Οι εταιρείε ε, υποστηρίζουν κάποια μεταπτυχιακά διδακτορικά προγράμματα για να λάβουν πόρου. Θα πρέπει όμω να γίνει κατανοητό το εξή. Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων μπορεί να επεκταθεί και σε άλλου τομεί. Οι εταιρείε μπορούν να συμμετάσχουν παραδείγματο χάρη και στη σύνταξη, στην κατάρτιση τη διδακτέας ύλη των πανεπιστημίων, στην κατάρτιση ίσω των ε, καθηγητών και να οργανώνουν και κάποιε περιόδου άσκηση ενδεχομένω. Θα μπορούσε να είναι ευεργετική λοιπόν η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων. Κατά τη σύνταξη τη έκθεσή μου ήρθα σε επαφή με εμπειρογνώμονε και από από τους δύο τομείς και από τι δύο πλευρέ. Και είδα ότι ένθεν κακήθεν συμφωνούν όλοι στο ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η σχέση και η συνεργασία μεταξύ πανεπιστήμιων και επιχειρήσεων. Ένα καθηγητή είπε ότι πέρασε πια η εποχή που τα πανεπιστήμια ήταν ερμητικά σφραγισμένα και κλειστά προς τον έξω κόσμο και ε, κεντρώνονταν μόνο στη θεωρία, ενώ ε, οι επιχειρήσεις αναπτύσσονταν από μόνες τους. Τώρα πλέον πρέπει να υπάρξει αλληλεξάρτηση διότι το μέλλον των πανεπιστημίων εξαρτάται από την ικανότητά του ε, να παράσχουν ανθρώπινο δυναμικό, στελεχικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που ενδιαφέρει του επιχειρηματίες είναι να έχουν ε, άτομα ε, εκπαιδευμένα, εξειδικευμένα, με γνώση τελευταία εχμής και με, τι κατάλληλε δεξιότητε. δεξιότητες. Πρέπει λοιπόν να γίνουν προσπάθειε και από τι δύο πλευρέ για ενίσχυση τη συνεργασία και βελτίωση του δυναμικού, των δυνατοτήτων. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην έκθεσή μου προσπαθώ να υπογραμμίσω τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενώ τις προσπάθειες αυτές διότι είμαι πεπισμένος ότι και οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι έχουν το συμφέρον να ε, βελτιωθεί αυτή η συνεργασία. πρέπει τα πανεπιστήμια ε, να παρέχουν πιο ε, καταρτισμένους εμπειρογνώμονες. Το πρόγραμμα 2020 αναφέρει και τη σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης, κάτι που απαιτεί τη στενότερη συνεργασία πανεπιστήμιων και επιχειρήσεων. Θέλω να προσθέσω ότι, όπως φάνηκε στις εκθέσεις, στην Ευρώπη ε, υστερούμε σε ό,τι αφορά την έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, σε ό,τι αφορά ε, τις επενδύσεις, ίσως κάτι 25% και περισσότερο. Τρεις τομείς ενίσχυσης της εργασίας θα ήθελα να αναφέρω. Διαβίου μάθηση είναι ένας τομέας. Εφιστώ την προσοχή σας στη σημασία της επιμόρφωσης, ε, της επανεκπαίδευσης. Θα πρέπει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνεργάζονται για τη χαρτογράφηση των αναγκών είναι σημαντικό να τονίσουμε και να παράσχουμε ευρύτερη πρόσβαση ε, στα πανεπιστήμια. Ε, η εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να βελτιωθεί. Όσοι δηλαδή ενήλικε θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, ε, θα πρέπει να τους δίνεται αυτή τη δυνατότητα και λαμβανομένου υπόψη και των δημογραφικών αλλαγών θα πρέπει να υπάρχει επίσης και ένα σύστημα παρακολούθησης ε, των αποφύτων και τη εξελίξή του τους ε, μετά στη σταδιοδρομία τους. Να υπάρχει και μια ανατροφοδότηση ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσον το πρόγραμμα σπουδών ε, συνάδει με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έχω διατυπώσει προτάσεις και για την κινητικότητα. Η κινητικότητα είναι ο ακρογωνίος λίθος της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής Μπορεί κανείς να μιλά για κινητικότητα σπουδαστών μεταξύ των χωρών μελών, αλλά μπορεί να ε, μιλήσει κανείς και για κινητικότητα μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, πιο καλά οργανωμένη και συντονισμένη συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων. Αυτού του είδους η κινητικότητα δεν έχει αναφερθεί τόσο πολύ και δεν είναι θέμα τόσο πόρων όσο θέμα οργάνωσης. Επίσης, προτείνω και οι τρίτες χώρες ε, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία ώστε να μπορούν τις χώρες αυτές ε, να εκπαιδεύονται εμπειρογνώμονες που θα είναι εξοικειωμένοι με τις ευρωπαϊκές μεθόδους και έπειτα να επιστρέφουν στη χώρα τους και να μπορούν να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες ε, να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτές τις χώρες. Ήρθα σε επαφή με διευθυντές, με μάνατζερ εταιριών, οι οποίοι ε, υποστήριξαν την ιδέα αυτή. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι το σύστημα ε, σταζιέρ των ε, μαθητευόμενων, των ασκούμενων. Έχουμε τα προγράμματα Erasmus, Leonardo. Είναι εξαιρετικέ δυνατότητε ενίσχυση αυτού του προγράμματο, αυτή τη σα. Διότι παρέχει πολύ σημαντική εμπειρία στου φοιτητέ που του βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα την αγορά εργασία και του παρέχει κίνητρα για περαιτέρω εκπαίδευση. Και στη διδακτή αίλη θα πρέπει να περιλαμβάνονται επιχειρηματικέ δεξιότητε και ικανότητε που μπορούν να βοηθήσουν του νέου αποφύτου να ξεκινήσουν τη δική του επιχείρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο της έκθεσής μου τονίζω τη σημασία των ε, βέλτιστων και αποδεδειγμένα καλών ε, πρακτικών. Σε κάποιους επαγγελματικούς τομείς ε, έχουν υπάρξει εδώ και καιρό κάποια προγράμματα τα οποία βασίζονται στη συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Αυτή λοιπόν η δέσμη γνώσης πρέπει να αξιοποιηθεί. Παραδείγματο χάρη, στο σελίδε στο διαδίκτυο Κυρία Πρόεδρε, σίγουρα είναι κατανοητό ότι όλα αυτά ίσως να αντιστοιχούν σε έναν ιδεατό κόσμο που οι φοιτητές γνωρίζουν ε, τι ε, πρέπει να επιτύχουν και πώς μπορούν να προοδεύσουν. Ο κόσμος όμως είναι πιο πολύπλοκος στην πραγματικότητα. Χρειάζεται χρηματοδότηση, ιδιωτικό κεφάλαιο, υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις, πρόσβαση στην εκπαίδευση, αναγνώριση, αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων σπουδών κτλ. Και αυτοί, αυτές οι πτυχές πρέπει να συμπεριληφθούν. Εγώ προσπάθησα στον πρώτο γύρο των συζητήσεων ε, άκουσα κάποιες προτάσεις και προσπάθησα να τις συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Τώρα θα γίνει μια συζήτηση που είμαι βέβαιος ότι θα συνεισφέρει και στη βελτίωση του κειμένου. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για την προσοχή και για τη δυνατότητα που μου δώσα να μιλήσω. Ευχαριστώ πάλι. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ριέρα Μαδουρέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πακ. Καταρχάς να πω ότι αποτελεί μεγάλη χαρά για μένα το γεγονός ότι μπορώ να συμμετάσχω στην ακρόαση αυτή της Επιτροπής ε, ε, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για ένα θέμα που όπως και εσείς εξηγήσατε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ενδιαφέρον και για την Κομισιόν Ήτρε. Σήμερα ψηφίστηκε η γνωμοδότησή μου στο, στην πρωινή συνεδρίαση. Η Επιτροπή Ήτρε δεν είναι μεν αρμόδια για θέματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά είναι αρμόδια για θέματα έρευνας. Και όπως γνωρίζετε, περίπου το 60% της έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται στα πανεπιστήμια. Επιπλέον, η Επιτροπή μας είναι αρμόδια και για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Επομένως, η Επιτροπή όπως είπατε και εσείς, έχει πολλά να πει σε ό,τι αφορά τη βελτίωση, την αύξηση, την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και το πώς μπορεί να γίνει αυτό. έρευνα και καινοτομία, αυτό το δίπτυχο έχουν πολλά ε, να συνεισφέρουν σε αυτή την πρόθεση, αυτό το διάλογο. Νομίζω ότι αυτό το διάλογο τον αναλύσαμε ε, και από τις δύο πλευρές και από τα δύο πρίσματα, δηλαδή και από την πλευρά των πανεπιστήμιων και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Σε αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου θα ήθελα απλά να σας ε, μεταφέρω κάποιες ιδέες ε, που ήταν αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαμε στην Επιτροπή Ήτρε και τις οποίες θέλω να συμπεριλάβω στην εκθεσή Πρέπει να σας πω ότι ορισμένες από αυτές τις ιδέες, πολλές από αυτές τις ιδέες, έχουν ήδη επισημανθεί από τους προλαλήσαντες Επομένως, απομένει να πω ότι συμφωνώ κατ' ουσίαν με όλα όσα υπόθηκαν, με όλες τις απόψεις που ακούστηκαν και θα ήθελα να αναφέρω απλά κάποιες ιδέες που δεν αναφέρθηκαν ακόμη και να τονίσω κάποιες άλλες από αυτές που ακούστηκαν ήδη. Πρώτη ιδέα είναι πολύ σημαντικό ο διάλογο αυτό μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων να είναι αμφίδρομο. Ε, δηλαδή να γίνεται και από την πλευρά τη ζήτηση και από την πλευρά τη προσφορά. Τι εννοώ. Αυτό ο διάλογο δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη διείσδυση τη επιχειρηματική κουλτούρα και νοοτροπία στο πανεπιστήμιο δηλαδή επιχειρηματικό πανεπιστήμιο αν θέλετε, θα πρέπει να οδηγήσει και στην ε, εισαγωγή της νοοτροπίας στις γνώσεις της επιχειρήσης πιο επιστημονικές επιχειρήσεις δηλαδή θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε αυτό. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν κατά την άποψή μα, σε ό,τι αφορά τη ζήτηση τα πανεπιστήμια, γιατί το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, αυτό τα πανεπιστήμια πάνω απ' όλα θα πρέπει να κάνουν μια καλή διάγνωση των ισχυρών τους σημείων στην εκπαίδευση, στην έρευνα και επίσης ποια είναι η σχέση των ισχυρών αυτών σημείων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Βέβαια, δεν θα πρέπει να λησμονούν τα πανεπιστήμια τον θεμελιώδη εκπαιδευτικό τους ρόλο, διότι το πρώτο βήμα για την επιτυχία και σε ό,τι αφορά δηλαδή και τη μεταφορά τεχνολογίας και τη σχέση με τις επιχειρήσεις είναι τα πανεπιστήμια να συνεισφέρουν στην αγορά εργασίας προσωπικό ε, υπαλλήλους εργαζόμενους με καλή εκπαίδευση, καλά προετοιμασμένους για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα με βάση τις γνώσεις και με βάση την αριστεία. Από την πλευρά της συζήτηση θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιώσουν ε, την ικανότητα απορρόφησης χρήσης και μετασχηματισμού των γνώσεων που παράγουν τα πανεπιστήμια στηρίζοντα, συμμετέχοντα σε ερευνητικά καθήκοντα και συμμετέχοντα ενεργά στα μεταπτυχιακά, στα διδακτορικά προγράμματα, όπω είπατε, στι υποτροφίε, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και ε, στην ε, πρόσληψη ερευνητών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την πρόθεση αυτή τη ε, αμφίδρομη σχέση, όπω είπα. Παραδείγματο χάρη, τεχνολογικέ πλατφόρμε, ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων ε, ε, κυρίως σε σχέση με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς και την έρευνα και όπως γίνεται και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο υπάρχουν κάποιες τεχνολογικές πλατφόρμες που όταν οριμάσουν μπορούν με φυσικό τρόπο να καταλήξουν σε συμπράξεις δημόσιου και δοτορικού τομέα όπως τα GTIs που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Στην έκθεση θελήσαμε επίσης να τονίσουμε ε, τον ε, ε, στόχο αυτό της σχέσης και της συνεργασίας δημόσιου ιδιωτικού τομέα γιατί θα είναι αμοιβαίως επωφελής και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, το Ευρωπαϊκό Τεχνολογίας ε, και Καινοτομίας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αρμοδιότητα της Επιτρόπου για την εκπαίδευση. Βέβαια και η Επιτροπή Ήτρε θα ήθελε να βλέπει κάποια μέλη του Ινστιτούτου αυτού, η IT και στην Επιτροπή μα. Να μην έρχονται μόνο στην Επιτροπή Πολιτισμού που είναι καθήλυνα, θέλω να έρχονται και στην Επιτροπή Ήτρε. Το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι το εξή. Συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες μορφές συνεργασίας για την πρόθεση αυτού του διαλόγου Αυτές οι μορφές όμως συνεργασίας, ε, σύνδεσης, εταιρικής σχέσης θα πρέπει να είναι δομημένες, καλά διαρθρωμένες. Ε, στο έγγραφο της Επιτροπής γίνεται λόγος για διαρθρωμένες, δομημένες μορφές. Είναι ένα ε, επίμαχο σημείο, διότι έχουν γίνει έρευνες και μελέτες από διάφορους εμπειρογνώμονες που θεωρούν ότι πιο αποδοτική μορφή αυτή τη στιγμή σχέσης είναι σε επίπεδο προσωπικών επαφών μέσω εκδόσεων, μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια, σε συνέδρια ή μέσω της παροχής ε, υπηρεσιών ε, και έρευνας ε, στο πλαίσιο συμβάσεων. Πρέπει δηλαδή να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι δομημένες μορφές μπορεί να είναι κάποτε υπερβολικά άκαμπτες και όχι τόσο ευέλικτες όσο οι μορφές που προανέφερα. Και επίσης θέλω να πω ότι και τα πανεπιστήμια δεν θα πρέπει να ξεχνούν δύο σημαντικές τους ε, ε, αποστολές που είναι η έρευνα και η εκπαίδευση και να περιορίζονται μόνο στην παραγωγή καινοτομίας. Ελπίζω να μην δημιουργηθούν προβλήματα πρόσθετα αντί να αντιμετωπιστούν τα είδε φυστάμενα. Πρέπει να τονίσουμε το σημαντικότατο ρόλο της κινητικότητας, της κινητικότητας σπουδαστών και φοιτητών ε, και ερευνητών βέβαια. Όταν μιλάμε για κινητικότητα φοιτητών και ερευνητών, συχνά μιλάμε για κινητικότητα μεταξύ χωρών. Εγώ θεωρώ σημαντικό να τονίσουμε, και αυτό γίνεται και στην έκθεσή μου, την κινητικότητα μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Και έρχομαι στο τρίτο σημείο το οποίο ήθελα να σας αναφέρω. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή και τα κρατημέλη θα πρέπει το νομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο να το αναθεωρήσουν για να ε, μην υπάρχουν φραγμοί στην κινητικότητα αυτή. Για μια ε, φορά επιτέλους να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια ενιαία αγορά ερευνητών ε, και βιομηχανική, συγγνώμη και διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης θα πρέπει να δοθούν κίνητρα Στι επιχειρήσεις με την άρση των ε, διοικητικών φραγμών. Και επίσης θα πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί που δίνουν περισσότερα κίνητρα και στα πανεπιστήμια. Και θα πρέπει βέβαια τα πανεπιστήμια να έχουν πλέον το κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά εν γέννη τη χρηματοδότηση, θα ήθελα να σημειώσω όχι μόνο το ρόλο των ε, κυβερνητικών οργανισμών και των επιχειρήσεων και ειδικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και ολοκληρώνοντας, τέταρτο σημείο, να επαναλάβω κάτι που υπόθηκε ήδη, ότι το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον διάλογο μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, μετά από τρία χρόνια λειτουργίας ε, απόρρια του έργου του είναι αυτή η έκθεση. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για την αντιτικοποίηση της συνεργασίας και του διαλόγου ε, μεταξύ πανεπιστημίων επιστημίων και επιχειρήσεων. Νομίζω ότι η εντατικοποίηση του διαλόγου είναι πάρα πολύ σημαντική για να ενισχυθεί το τρίγωνο της ε, γνώσης. Αυτό θα είναι προς αμοιβαίο όφελος, δηλαδή προς όφελος και των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Γνώση, networking, διαδικτύωση, ανταγωνιστικότητα επίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζουμε επίσης ότι είναι πολύ καλή ιδέα που εξέφρασε η πρώτη ομιλήτρια στα επίπεδα των κρατών μελών και στο περιφερειακό επίπεδο να υπάρξει μια επέκταση αυτού του προγράμματος αλλά βέβαια θα πρέπει τα πανεπιστήμια να παραμείνουν αυτόνομα και δημόσια. Και στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου δεν θα πρέπει απλά μόνο να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας όπως ε, είπε ο εισηγητής αλλά θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν οι καλύτερες δυνατές πολιτικές και τα καλύτερα δυνατά μέσα, εργαλεία που υπάρχουν σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να έχουμε τη μεταφορά γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, διότι τελικά όπως προείπα τα πανεπιστήμια βλέπουμε να αντιδρούν πλέον θετικά ε, στα εφιστάμενα κίνητρα, στα περιφερειακά, εθνικά και κοινοτικά ε, προγράμματα για την ανάπτυξη πολιτικών συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σας αναφέρω μια ιδέα την οποία αναφέρει η Κομισιόν στον έγγραφό της και την οποία ανέφεραν και ορισμένοι από τους προλαλήσαντες και την οποία εγώ θεωρώ πολύ σημαντική αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να δώσουμε μια δυνατή όθεση στην εργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Ε, σε καιρού ε, οικονομική ύφεση, όταν δηλαδή οι φοιτητέ δυσκολεύονται περισσότερο από άλλε εποχέ για να βρουν δουλειά και όταν ε, οι επιχειρήσει αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερε ανταγωνιστικέ πιέσει, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Διότι αυτή η συνεργασία έχει προστιθέμενη οικονομική και κοινωνική αξία. Και αυτή η σχέση γίνεται όλο και πιο αναγκαία και αποτελεί όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα. Και στο ίδιο πλαίσιο θέλω να τονίσω πόσο εύστοχη και επίκαιρη είναι αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαντουρέλ. Δεν έρχεστε σε αντίθεση μεταξύ σας, αλλά λίγο συμπληρώνεστε. Αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια έχουν κοινού στόχου προς το συμφέρον των φοιτητών. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε καλό δρόμο. Η Ένωση προσφέρει μια πλατφόρμα όπου οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνδέσεις μπορούν και πρέπει να γίνουν. Ελπίζω να υπάρξει συνειδητοποίηση αυτών των ευκαιριών και ευχαριστούμε την Κομισιόν που μας κάνει αυτή την πρόταση η κυρία Μπερνάντο Ντεκβέρος, αν θέλει να προσθέσει κάτι στι δύο αυτέ παρεμβάσει, τώρα είναι η στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ε, όταν μίλησα για εισηγήτρια ή εισηγητή ε, στα ισπανικά η λέξη που χρησιμοποίησα δεν αναφέρεται μόνο σε εισηγητή έκθεση στο κοινοβουλίο αλλά και σε κάποιον που παρουσιάζει μια εισήγηση ε, ζητώ συγγνώμη. Να απαντήσω τώρα στον συντάκτη γνωμοδότηση, στον κύριο Πάλι Σμιθ. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, φυσικά και συμφωνούμε πλήρως με την έκθεση του κυρίου Πάλι Σμιθ που συμφωνεί απόλυτα με τις βασικές γραμμές πολιτικής της Κομισιόν και τα θεματικά φόρα και τις τελευταίες σκέψεις και προβληματισμού. Συμφωνούμε και με τη διάγνωση την οποία προέβη. Είναι σαφές ότι μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων, ε, το να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία και προσοχή και στις ανάγκες της αγοράς θα είναι επωφελή όχι μόνο των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, αλλά τελικά επωφελή του ίδιου του πολίτη και επίσης το γεγονός ότι θα είναι πιο ανοιχτά τα πανεπιστήμια ε, του πολίτες, αυτό θα συνιστά και έναν παράγοντα ανάπτυξη. Αυτό μα βρίσκει σύμφωνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί υπέρ διαφόρων μέτρων. Πρώτα απ' όλα σκεφτόμαστε πώ μπορούμε να αναλύσουμε νέα θέματα, θέματα τα οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα να θίξουμε μέχρι στιγμή. Όπω παραδείγματο χάρη μικρομεσαίε επιχειρήσει που αναφέρατε, περιφερειακή συνεργασία, καινοτομία, ε, επιχειρηματικότητα και ίσως ένα τελευταίο θέμα συνεργασία ε, πανεπιστημίων επιχειρήσεων στις κοινωνικές επιστήμες. Αυτά τα επεξεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτόν τον καιρό. Όπως γνωρίζετε όλα τα αποτελέσματα των διαφόρων βημάτων συζήτησης ε, ε, θα τα δείτε στις ιστοσελίδες των εταιρικών σχέσεων και έχουμε και δύο μεγάλα ανοιχτά θέματα. Το πρώτο είναι η μελέτη των καλών πρακτικών που θα δρομολογηθεί όπως γνωρίζετε το Μάρτιο και που έχει ως στόχο τον εντοπισμό 30 καλών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον η εικονική πλατφόρμα που γίνεται αυτή τη στιγμή μελέτη σκοπιμότητας ε, για να δούμε κατά πόσον μπορεί να υλοποιηθεί και ίσως μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε σε πραγματικό χρόνο μια συνέχιση του διαλόγου των ε, πλεκομένων φορέων χωρίς να χρειάζεται να συναντιόνται ε, αυτοί οι άνθρωποι. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια από τα σχόλια της συντάκτρας γνωμοδότησης, τονίζοντας και δύο. Πρώτα απ' όλα για τον κύριο Σμίθ, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τους φραγμούς κατά της κινητικότητα. Συμφωνούμε απόλυτα και βέβαια για να γίνει αυτό θα πρέπει και οι ε, αρχές, οι δημόσιες αρχές ε, να ε, συνεισφέρουν δεν έχουμε μόνο το ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε και το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να προβλεφθούν περισσότερες δυνατότητες ε, πρακτικής άσκησης, περίοδου άσκησης ε, στις επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι το Εράσμος κάνει σημαντική δουλειά στον τομέα αυτό, αλλά δεν αρκεί, πρέπει να συνεχίσουμε. Και τέλος, όπως γνωρίζετε, εδώ και κάποιο καιρό ε, το ETF σε αυτό το θέμα ε, συνεργάζεται μαζί μας. Γίνεται μια ανάλυση των ε, συμπράξεων πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και συντονικέ χώρε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ΙΤΕΦ ε, είχε μια, ένα πρώτο βήμα συζήτηση το Δεκέμβριο, πολύ επιτυχημένο, 2 και 3 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, και εκ παραλίλου τότε και μαζί μας διεξαγόταν και μια μελέτη καλών πρακτικών. Όλες αυτές λοιπόν οι εργασίες μας, αυτά τα δύο ανοιχτά θέματα, σύντομα ελπίζω να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η δέσμη αυτή μας δίνει ιδιαίτερη όθηση. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και ερχόμαστε στο θέμα του απογεύματο. που ξεπερνάει τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προκλήσεις και απαντήσεις. Δεν είναι μόνο επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο. Χαίρομαι για το ότι χρειάστηκε να προσκαλέσουμε εμπειρογνώμονες στην ακρόση τον καθηγητή Ντόναλ Καπ, διευθυντή του Κέντρου Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κωνσταντσα από το Πανεπιστήμιο της Θαλάσσης στη Ρουμανία. Ο κύριος Καπ, καλώς ορίσατε. Καθηγητής Ρόμπερ Γκάμπριελ, πριν του Πανεπιστημίου του Πίτς στην Ουγγαρία. Η Πίτς είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα με την Έσεν και την Κωνσταντινούπολη φέτος. Φλόριαν Κάιζερ, εκπρόσωπος των φοιτητών από τη Γερμανία. Καθηγητή Χόουαρτ Νιούμπι, πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα θα έρθει η κυρία Έλεν Κλάρκ από την Lifelong Learning Policy εκ μέρους της Κομισιόν και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τζάβερ Γκοντζάλες Βέγκα που θα μιλήσει εκ μέρους του Συμβουλίου. Σας προτείνω το εξής, οργανωτικά. Ο κάθε εμπειρογνώμονας έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του να μιλήσει. Παρακαλώ μην τα ξεπερνάτε. Μετά θα τεθούν ερωτήσεις και απαντήσεις συνολικά 15 λεπτά. Και παρακαλώ τους συναδέφους να είναι λακωνικοί, να μένουν στο συγκεκριμένο ερώτημά τους, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία πολλοί βουλευτές να μιλήσουν. Και τέλος, θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν και τον εκπρόσωπο της, του Συμβουλίου. Έχουμε εδώ ένα έγγραφο όπως βλέπετε που είναι η θέση της ε, Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Ο συγητής, ο κύριος Φανέρσελ, είναι παρόν. Πάρα πολύ καλή δουλειά του συναδέλφου από την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή. Και μια τεχνική ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αυτή μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Γι' αυτό παρακαλώ όποιος μιλάει να ανοίγει το μικρόφωνο και με το που τελειώνει την ομιλία του να κλείνει το μικρόφωνο. Είναι εξίσου σημαντικό. Σε ζητάω συγγνώμη αν κάτι ξέχασα. Θα χρειαστεί να φύγω γιατί έχω μια ομάδα επισκεπτών από την εκλογική μου περιφέρεια. Πρέπει να τους συναντήσω, θα φύγω και παρακαλώ τον συνάδελφο Σόνι να αναλάβει την προεδρία στη θέση μου. arvoisa esitelmöitsijä hyvä και κύριοι, ευχαριστώ. Η δόκτωρ Ντόινα Κάρπ μπορεί να ξεκινήσει. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί βουλευτέ, παρά την την επιφαινόμενη αδράνεια, τα τελευταία 700 χρόνια τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν διατηρήσει την ανεξαρτησία τους. Και πολύ περισσότερο από το 18ο αιώνα και μετά και είναι πάντοτε σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Τον 20ο αιώνα μάλιστα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έγιναν πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού συστήματο, ενώ το, το εσωτερικό, η εσωτερική του οργάνωση μεταρρυθμίστηκε τελείως. Ε, οι παράγοντες και τα αίτια που καθόρισαν τις πανεπιστημιακές πολιτικές ε, ασχολήθηκαν και με την υποδοχή, τη διαφορετική υποδοχή των φοιτητών και με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Έτσι τα πανεπιστήμια κάποιες φορές ε, στη νέα τους ε, μορφή παρουσίασαν δυσκολίες. Δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν και χρειάστηκαν ε, εκβάθρων ε, μεταρρυθμίσεις. Και αυτό προκειμένου τα πανεπιστήμια να γίνουν ένας λειτουργικό θεσμός για, το νεό, για την ευρωπαϊκή νεολαία πανεπιστήμια λοιπόν δεν πρέπει να τα βλέπουμε ως ένα χώρο απομονωμένο πέραν του υπόλοιπου πολιτικού σκηνικού. Τον 21ο αιώνα τα πανεπιστήμια αναζητούν και οικονομικές λύσεις για να διατηρηθεί η δραστηριότητά τους, ενώ τα πράγματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και συνεχώς απαιτείται περαιτέρω επέκταση της δράσης τους η γενίκευση της ε, διδασκαλίας από την ελιτιστική εκπαίδευση προς την ε, διάδοσή της ε, έχει φτάσει πλέον και στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών μέσων. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πανεπιστήμια πλέον κρίνονται ανάλογα με την ε, μονομένη τους αξία. Ενώ ε, το ιδιαίτερο κύρος των καθηγητών πανεπιστημίων στην κοινωνία έχει μειωθεί. Ένα καθεστώς που ήταν αδιαμφισβήτητο επί αιώνες. Τα πανεπιστήμια στην κοινωνία της γνώσης. Η κοινωνία αυτή συσχετίζει τέσσερα ανεξάρτητα στοιχεία. Η παραγωγή της γνώσης είναι απαραίτητη για την επιστημονική έρευνα. Έπειτα, η μετάδοση της γνώσης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και κατά τρίτον, η διάδοση της γνώσης μέσω της τεχνολογίας, της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Τέταρτον, η αξιοποίηση της γνώσης μέσω της τεχνολογικής καινοτομία. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι γνώσεις βρίσκονται σε ένα στάδιο μεταξύ τη έρευνα, τη καινοτομία ε, και τη πρόοδου. Έτσι λοιπόν τα πανεπιστήμια κρατούν το κλειδί τη πρόοδου τη κοινωνία, βασισμένη στην γνώση. Επίση, τα πανεπιστήμια συνεισφέρουν στην υλοποίηση και άλλων στόχων τη στρατηγικής τη Λισαβόνα, όπω υπόθηκε και προηγουμένω, όπω η κοινωνική συνοχή ή η βελτίωση του γενικότερου μορφωτικού επίπεδου στην Ευρώπη οι τομείς όπου τα πανεπιστήμια ε, έχουν καθοριστικό ρόλο να διδραματίσουν είναι η επιστημονική έρευνα και η διάδοση των πορισμάτων της μέσω της συνεργασίας των βιομηχανιών ή μέσω των εταιρικών σχέσεων για σκοπούς έρευνας. Η αξιοποίηση των ερευνητών στα πανεπιστήμια αλλά και των εκπαιδευτών ή των καθηγητών για την προπανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι ε, σημαντικά στοιχεία. Δεν είναι όμως μόνο τα πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν ε, τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, αλλά και οι οργανώσεις, οι εμπορικές ενώσεις και οι επιχειρήσεις βεβαίως που έρχονται πλέον προς τον ακαδημαϊκό κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν τα αιτήματα και ανάγκες των ΜΕ να προσαρμόζονται στα αιτήματα και τις ανάγκες των ΔΕ ώστε οι κοινοί του στόχοι να επιδιώκονται με μια συμφωνία, με μια σύγκληση. Το σκηνικό, το ευρωπαϊκό σκηνικό των ανάπτωτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπω είναι οργανωμένο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, είναι αρκετά ετερογενέ ω προ την διοργάνωση των ιδρυμάτων, ω προ την χρηματοδότησή του και ω προ τι συνθήκε λειτουργία του. Αυτή η ετερογένεια ε, είναι χαρακτηριστική μεταξύ των χωρών λόγω των διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων και των διαφορετικών νομοθεσιών αλλά και εντός της κάθε μια χώρας αναλόγως ε, με την ανεξαρτησία του κάθε πανεπιστημίου ή με την ταχύτητα εξέλιξής του. Η διαδικασία της ε, Μπολόνια είναι μια σοβαρή προσπάθεια διοργάνωσης των πανεπιστημίων παρά την ε, διαφορά τους και τη διαφορετικότητά τους σε ένα πιο συνεκτικό και πιο ενιαίο ευρωπαϊκό σκηνικό. Η διοργάνωση των σπουδών σε τρεις βαθμίδες, ε, πρώτο πτυχίο, μάστερ και διδακτορικό, δίνει τη δυνατότητα ε, σε φοιτητέ να αποκτήσουν ε, βάσει ενό αριθμού σπουδών και ένα συγκεκριμένο δίπλωμα. Επίσης έχουμε και την ε, έννοια του στάζ, την πρακτική δηλαδή σε επιχειρήσεις που συμπληρώνει τη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών. Αυτή όμω η πρακτική κατάρτιση απαιτεί διαφορετική διοργάνωση των σπουδών στη διάρκεια του χρόνου. Έτσι χρησιμοποιείται αναλλαγή μεταξύ πρακτικών και τεχνικών σπουδών κάτι που υποχρέωσε την αλλαγή των ακαδημαϊκών προγραμμάτων των πανεπιστημίων, επιτρέποντα σε όσου εργάζονται να έρθουν και πάλι κοντά στα πανεπιστήμια, ακολουθώντα συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Δέκα χρόνια μετά την αρχή τη διαδικασία τη Μπολόνια, και με την μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων των, πανεπιστημίων και τη μετατροπή τους σε ενεργά και αντιδραστικά συστήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, έχουμε πλέον μια νέα γενιά καθηγητών, εκπαιδευτών ε, και υπευθύνων για την κατάρτιση, καθώς και νέες επαγγελματικές σχέσεις στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν τις επιτακτικές ανάγκες ε, που το δύσκολο περιβάλλον, το ασταθές περιβάλλον της εργασίας επιβάλλει. Έχει αλλάξει πλέον ο τόπος παραγωγής της γνώσης. Ε, επίκυνται και άλλες αλλαγές. Υπάρχει πιο στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και οικονομικού τομέα. Οι οργανώσεις, οι εμπορικές ενώσεις χρησιμοποιούν όλα τους τα μέσα για την παραγωγή γνώσης και έχουν διαφορετικέ προκλήσει μπροστά του, όπω την ανάγκη τη διαδίου κατάρτιση, προκειμένου να, να παραμείνουν ανταγωνιστικέ και αποδοτικέ μακροπρόθεσμα. Η ανάπτυξη τη γνώση ε, κατά τρόπο συστηματικό, η ενημέρωση για τα προϊόντα, τι διαδικασίε και τη διοργάνωση είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είναι το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να παραχθεί και άλλη γνώση για την διοργάνωση των επιχειρήσεων. Εξαιτίας αυτών των συνθήκων ο ακαδημαϊκός και επιχειρησιακός κόσμος έρχονται όλο και πιο κοντά και αλληλοσυμπληρώνονται. Ίσως ε, να καταλήξουν οι δύο αυτοί κόσμοι να κινούνται παράλληλα και σε συγχρονία τον 20ο και 21ο αιώνα. Ε, η, σταθερότητα, η γνωστή σταθερότητα έχει μεταβληθεί η ζήτηση καθορίζει την ε, δομή των πανεπιστημίων και όχι πλέον άλλες ε, πεπιθήσεις όπως οι θρησκευτικέ. Η διεπιστημονική κατάρτιση, η ανάγκη κάλυψης των θέσεων στην αγορά εργασίας, αυτή οι, αυτές οι τάσεις μαζί με, την, με το ασταθές περιβάλλον είναι σημαντικό οι οικονομίες εχμής, αλλά και όλοι οι οικονομικοί τομεί είναι τομεί που του αφορούν αυτέ οι αλλαγέ. Έτσι, όταν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητε επιχειρηματικότητα. Η αύξηση της ζήτησης για πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε όλους τους τομείς τι τελευταίες δεκαετίες καθώς δεν συνοδεύεται και από απαραίτητη αύξηση της γεννητικότητας Παρόλα αυτά, μας οδηγεί να θέσουμε μια σειρά από ερωτήματα. Τι να κάνουμε για να εκπαιδεύσουμε καθηγητές και εκπαιδευτές ποιότητας. Η ποιότητα ούτως ή άλλως πρέπει να συνδυαστεί και με την κατάλληλη διάρκεια. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε την αριστεία καθ' όλη αυτή τη διαδικασία και στη διδασκαλία και στην έρευνα. Οι αλλαγές αυτές έχουν επιταχυνθεί από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας, της έρευνας και της πληροφορίας. Η στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων, ερευνητικών Ινστιτούτων, είναι άκρο αναγκαία. Μέρος της χρηματοδότησης αποκτάται τόσο ή άλλως κατά τρόπο ανταγωνιστικό. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν μπορεί να κρατήσει και να κινητοποιήσει τους καλύτερα καταρτισμένους και πιο πρικισμένους καθηγητές ε, στον χώρο τον ακαδημαϊκό. Επίσης, οι Ευρωπαίοι φοιτητές μετά το τέλος των σπουδών τους μπορεί να παραμείνουν στην Ευρώπη, τουλάχιστον ή άριστοι. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε στην Ευρώπη πανεπιστημιακούς πόλους, ακαδημαϊκούς πόλους έλξης για τους φοιτητές που να είναι πολύ ισχυροί. κατά παραδοσιακό τρόπο τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ασχολούνται με τη διάδοση των ερευνητικών πορισμάτων. Όμως υπάρχουν και άλλα σημεία που μπορούν να γίνουν ε, να γίνει έρευνα στις επιχειρήσεις, ε, στις εταιρείες, όπου πολλές φορές οι εργαζόμενοι είναι επαγγελματίες με ψηλά προσόντα, παράγουν γνώση και μπορούν να χρησιμοποιήσουν για συγκεκριμένους σκοπούς τη γνώση που παράγουν. Υπάρχει λοιπόν μια τάση τα πορίσματα αυτά τα ερευνητικά να συμπεριληφθούν στη γενικότερη έννοια τη γνώση όπω ορίζεται στα πανεπιστημία. Και έτσι βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα χώρο σύγκλησης και ανταγωνισμού μεταξύ πανεπιστημίων και επιχείρησης. Η αναδιοργάνωση λοιπόν της ε, γνώσης και η ανάγκη αυτή ε, φαίνεται να παρουσιάζει δύο τάσεις. Περισσότερη ειδίκευση και επικάλυψη μεταξύ έρευνας στην εκπαίδευση και έρευνα στις επιχειρήσεις και από την άλλη η ανάγκη προσαρμογής προσαρμογή στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών. Βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρία διαφορετικά κινήματα που εξελίσσονται παράλληλα, αλλά είναι πτυχέ της ίδιας διαδικασία. Ο ευρωπαϊκό χώρο τη ενότητας εκπαίδευση, ο ρόλο τη ε, κατάρτιση των ενηλίκων, τη διαβίου μάθηση δηλαδή, και οι πτυχέ αυτέ θα είναι η επόμενη αποστολή που θα αναλάβουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τις ερχόμενες δεκαετίες. Να αναφέρω εδώ και μια σημαντική λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης ε, μια λειτουργία την οποία σπάνια αναφέρουμε. Δηλαδή να διασφαλίσει μέσω υψηλών προσόντων προσωπικού την ε, εκπαίδευση, των κύκλο μαθημάτων. Βασιζόμαστε εδώ στην ε, θεωρία ότι οι γνώσεις των μελλοντικών γενιών θα είναι καθοριστική σημασία για το μέλλον. Όμως την εκπαίδευση αυτή ποιοι θα την παρέχουν. Πρέπει να είναι καθηγητέ κατά την παραδοσιακή έννοια, να ανήκουν σε αυτή την κοινωνική κατηγορία. Όμω, οι καθηγητέ τη Ευρώπη θα πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου ούτω ή άλλω, αλλά με πολύ συγκεκριμένε ικανότητε και δεξιότητε για τον 21ο αιώνα. Δηλαδή, να γνωρίζουν τον επιστημονικό του κλάδο, να είναι σε θέση να οργανώσουν την εκπαίδευση, να δημιουργήσουν ευκαιρίε για του φοιτητέ και επιπλέον να παρακολουθήσουν τις πρόοδους των φοιτητών Δηλαδή να μπορούν να διαχειριστούν ομάδες ε, με διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις, με διαφορετικές ανάγκες και να σεβαστούν και τη δίψα και των φοιτητών. Θα πρέπει οι φοιτητές να μπορούν να οργαστούν συλλογικά. Οι γονείς να ασχοληθούν με τα προβλήματα του πανεπιστημίου, οι νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα, καθώς και νέες παιδαγωγικές μέθοδοι να αξιοποιηθούν. Και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον δεοντολογικά άρτιο. Στο θα πρέπει να σκεφτούμε επί της ουσίας πώς πρέπει να έχουμε μια παιδαγωγική μέθοδο, μια δοντολογία εύστοχες. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε από τώρα. Από τώρα να αρχίσουν να μας απασχολούν. Οι σημερινοί φοιτητέ θα είναι κατά αυτόν τον τρόπο σε θέση αύριο να εκπαιδεύσουν άλλους φοιτητέ και να αναλάβουν την ευθύνη και τις ε, απαραίτητες δεξιότητες για να γίνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες. Εν am κατακλείδη ήθελα να αναφέρω μια κινέζικη παροιμία. Πολύ εύστοχη εδώ που μιλά για την εκπαίδευση στο μέλλον. Και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την προσκλήση. Paljon kiitoksia, tohtori Doina Karp, ja seuraavaksi σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τον λόγο έχει ο Δόκτωρ Γκάμπριλ για 10 λεπτά. Κύριε καθηγητά, αν είστε έτοιμος μπορείτε να αρχίσετε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, θα τοποθετηθώ κάπως διαφορετικά σε σχέση με τον προηγούμενο μιλητή. Θα σας πω τις απόψεις μου και θα κάνω και μερικά ερωτήματα, όπως ζήτησε η κυρία Πάκ στην εισαγωγή της. Χρειαζόμαστε ερωτήσεις για να έχουμε απαντήσεις. Θα κάνω ερωτήματα, θα υποβάλω ερωτήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επικεφαλής των πανεπιστημίων. Καταρχήν, ποια είναι η προοπτική μου. Είμαι επικεφαλής πρίτανης του Πανεπιστημίου που είναι από πιο παλιά πανεπιστήμια και επιχειρήσεις θα έλεγα. 30.000 φοιτητές έχουμε είμαστε η πιο μεγάλη μονάδα. Θεωρώ το Πανεπιστήμιό μου ως μια επιχείρηση και αντιμετωπίζω το έργο μου ως επιχειρηματίας σε θέματα μεταφοράς επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογίας. Σύντομα θα αναφερθώ στα εξής δύο τεινά στις σχέσεις επιχειρήσεων πανεπιστημίων. Το είναι ο ρόλος των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην κατάρτιση προκειμένου να υπάρξει ένα κατάλληλο εργατικό δυναμικό για την αγορά. Αυτό είναι από τα βασικά ερωτήματα που μας τίθεται από τις επιχειρήσεις τις ίδιες. Και το δεύτερο είναι η συμβολή των πανεπιστημίων στην έρευνα και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σας δείχνω ένα διάγραμμα όπου βλέπετε μερικά βιβλία και τίτλους για τα πανεπιστήμια είναι μεγάλη πρόκληση πώς θα επιλέξουμε ένα βιβλίο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα βιβλίο για να διδάξουμε τους φοιτητές μας ένα εγχειρίδιο. Βέβαια η απάντησή μου είναι όχι μόνο ένα εγχειρίδιο. Η σωστή λύση είναι ένας συνδυασμός πολλών εγχειρίδιων. Καταρχήν η ευθύνη των πανεπιστημιακών. Εδώ υπάρχουν δύο βασικοί φορείς και εφαίροι. Είναι η, η, η πολύ σημαντική πανεπιστημιακή που κάνουν την έρευνα και άλλη είναι η διοικητική των πανεπιστημίων. Διαφορετικός ο ρόλος του καθενός στις σχέσεις επιχειρήσεων πανεπιστημίων. Ο βασικός ρόλος των πανεπιστημιακών είναι να ορίσουν ε, σύγχρονη διδακτέα ύλη για τους φοιτητές και να ενημερώνουν, να φρεσκάρουν τις επιστημονικές γνώσεις. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τους φοιτητές. Η διαβίω ανάπτυξη, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καθημερινή μας ζωή. Το τονίζω αυτό με πολλές εικόνες, όπως βλέπετε. Βλέπετε ένα σκάνινγκ εδώ του εγκεφάλου που μας δείχνει τρεις περιοχές. Πρώτον, χρειαζόμαστε θεωρητική γνώση των πραγμάτων για το οποίο μιλάει κανείς ή ερευνά κανείς. Το δεύτερο είναι χρειάζεται συνδυασμός δεξιοτήτων για τη σύγχρονη έρευνα και το τρίτο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα από τη σκοπιά της ψηλής τεχνολογίας. Ένα να λείπει, κάτι δεν πάει καλά. Ε, βλέπετε πως αυτές οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις άγγελο συμπληρώνονται ή άγγελο επικαλύπτονται. Χρειαζόμαστε τις ικανότητες αυτές. Δηλαδή υψηλή τεχνολογία, ε, δεξιότητες του μυαλού προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας. Ο δεύτερος ρόλος είναι να χαρακτεί η ερευνητική κατεύθυνση στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι πρωτεύουσα σημασία σήμερα, διότι η έρευνα είναι ένα πολύ ευρύ τομέα. Οι δυνατότητε είναι πάρα πολλέ αυτή τη στιγμή για έρευνα και χρειάζεται επιλογή προκειμένου να πετύχουμε γρήγορα τις καινοτομίες που θέλουμε. Στα πανεπιστήμια λοιπόν αυτές οι δύο ομάδες, οι διοικητικοί και οι ερευνητές, έχουν λίγο διαφορετικούς ρόλους. και μερικές φορές έρχονται και σε αντίθεση η μία ομάδα με την άλλη. Αλλά και οι δυο χρειάζονται προκειμένου να έχουμε ε, ένα αναπτυγμένο ερευνητικό και αναπτυξιακό δυναμικό στα πανεπιστήμια. Επίσης πρέπει να υπάρχει και ροή κονδυλίων και από την κυβέρνηση και από την Ένωση. Αυτό το φροντίζουν οι διοικητικοί, αλλά αν οι καθαρά πανεπιστημιακοί ερευνητές και λοιπά δεν παράγουν αποτελέσματα, τελικά δεν θα έχουμε ένα βιώσιμο πανεπιστήμιο. Άλλο μεγάλο θέμα είναι ποια είναι η σχέση του πανεπιστημίου με την κοινωνία. Το πανεπιστήμιο πρέπει να εξυπηρετεί την κοινωνία, πρέπει να είναι πιο ευέλικτο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Πρέπει να είναι αυτοϋποστηριζόμενο και να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και της έρευνας και της διδασκαλίας. Ήδη ακούσαμε ότι ασκούνται επικρίσεις σχετικά με τα, τα αιτήματα της οικονομίας και το τι δίνει το Πανεπιστήμιο. Ότι δεν υπάρχει μία πλήρης συμφωνία μεταξύ των δεξιοτήτων που δίνουν τα πανεπιστήμια και από την άλλη μια πλήρη συμφωνια μεταξυ των δεξιοτητων που δινουν τα πανεπιστημια και απο την αλλη μια ελλειψη σε επιστημονικές δεξιότητες. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και η Ένωση και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ξανασκεφτεί την πολιτική τους για το θέμα αυτό. Αν λυθεί το μικρό αυτό πρόβλημα που βλέπετε στην οθόνη αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε κανείς να πάρει ένα διδακτορικό. λύνοντα το πρόβλημα αυτό και μόνο. Βέβαια υπάρχουν πολλά αίτια για την κατάσταση αυτή. Το ένα είναι το ότι η επιστήμη δεν είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Πριν από 30-40 χρόνια οι θετικέ επιστήμε ήταν πολύ πιο δημοφιλεί στα σχολεία από ό,τι σήμερα. Θεωρείται δύσκολο να μάθει κανεί θετικέ επιστήμε στα λύκεια, στα πανεπιστήμια. Αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε. Να γυρίσουμε στην εκλαϊκευμένη επιστήμη και να καταφέρουμε να τραβάμε περισσότερο κόσμο στις θετικές επιστήμες. Δεύτερο είναι στις θετικές επιστήμες, στα πανεπιστήμια, η μισθή είναι πιο χαμηλή από τις επιχειρήσεις. Εδώ μπορεί να βοηθήσει η νομοθεσία. Δεν γίνεται μόνο με προσφορά και ζήτηση αυτό. Χρειάζεται ρύθμιση, μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδο ένωσης, σε τοπικό επίπεδο, πάντως πρέπει να υπάρξει ρύθμιση γι' αυτό. Αν θέλετε να γυρίσουμε μερικοί στις, ε, στο χώρο των θετικών επιστημών, πολυτεχνία κλπ. Και το τρίτο είναι ότι δεν υπάρχει feedback, δεν υπάρχει ανάδραση εκ μέρους της αγοράς εργασίας σχετικά με το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Τα πανεπιστήμια παίρνουν φοιτητέ χωρίς να έχουν αυτό το feedback από την κοινωνία και από τις επιχειρήσεις. Θα μπορούσα να πω και δύο λόγια επίσης για την διαβίω ε, εκπαίδευση, lifelong. Πολύ δύσκολο και το θέμα αυτό και αφορά ε, τι θα πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στους νέους φοιτητές, να στηριζόμαστε και σε άτομα που είναι πιο μεγάλη σε ηλικία αλλά θέλουν να ξαναμπούν μέσα στο σύστημα το εκπαιδευτικό. Γιατί αυτό αφορά και την κατανομή των ηλικιών στην Ευρώπη αλλά αφορά και προβλήματα που οφείλονται στη βασική εκπαίδευση. Δηλαδή είναι δύσκολο να ε, καλέσουμε άτομα στην, ε, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση αν είναι σχεδόν αναλφάβητοι. Θα πρέπει να ξαναδούμε δηλαδή και τη βασική εκπαίδευση, αν ο στόχο μα είναι τα πανεπιστήμια, και τη βασική την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Φυσικά μετά χρειάζονται γλώσσε, βασικέ γνώσει Όλα αυτά είναι θετικά. Υπάρχει και μια μεγάλη πρόκληση όμως για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Το ECTS, το σύστημα μεταφοράς των βαθμών, δεν ισχύει απόλυτα. Συνήθως όταν κάποιος φοιτής με ρωτάει τι να κάνω σχετικά με την κινητικότητα, εγώ το συμβουλεύω να κινηθεί μεταξύ των κύκλων, όχι μέσα σε ένα κύκλο. Γιατί ένας κύκλος σπουδών είναι σχετικά σύντομος και δεν βοηθάει προκειμένου να αποκτήσει την εμπειρία αυτή που χρειάζεται μέσα σε δύο ή τρία χρόνια. Καλύτερα να κινηθεί μεταξύ των κύκλων όταν θα πέρασει Φερπίν προς το Μάσταρ. Και μία τελευταία διαφάνεια για την έρευνα και ανάπτυξη και την, τη δυνατότητα δίνει στις θετικές επιστήμες. Ένα μεγάλο δίλημα για τους επιστήμονες. Είναι γνωστό δίλημα για τους επιστήμονες. Ένας επιστήμονας ψηλού πρέπει να δημοσιεύει κάπως να δημοσιεύει το χρόνο. Αν δημοσιεύσει όμως συμβαίνει δύο τινά. Πρώτον, δεν έχει χρόνο για να κάνει έρευνα ο επιστήμονας και μερικές φορές τα συμβόλαια σε απαγορεύουν να δημοσιεύσει τα πορίσματα αυτά. Μεγάλο δίλημα αυτό για τους επιστήμονες. Έπειτα έχουμε τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να είναι ένα θέμα που να αφορά και τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια. Το ιδιώδες θα ήταν οι ερευνητές, τα πανεπιστήμια και επιχειρήσεις από κοινού να δουλεύουν. Γιατί εκεί τίθεται θέμα εμπιστοσύνη μεταξύ και των επιχειρήσεων και των επιμέρους ερευνητών και των πανεπιστημίων. Αυτό η τριμερή σύνθεση, η τριμερή συμμετοχή θα έδινε τα άριστα αποτελέσματα κατά τη γνώμη μου. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο μας, με τελικά αποτελέσματα τον Αύγουστο του 2011. Ελπίζουμε να ξεκινήσει μια νέα χρονιά και μια νέα περίοδος πραγματικά για το Πανεπιστήμιό μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε καθηγητά Γκάμπριελ. Και τώρα ο κύριος Κάιζερ. Για 10 λεπτά έχετε το λόγο. Zunächst mal vielen Dank für die Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα και στους φοιτητές να μιλήσουν για το μέλλον των πανεπιστημίων, διότι είναι ένα θέμα που μας ε, απασχολεί καθημερινώς. Επέλεξα κάτι πολύ συγκεκριμένο, τη διαδικασία της Μπολόνια, διότι τίθενται σημαντικά ζητήματα τα οποία στο μέλλον θα επιμείνουν τέλος πάντων θα δώσουν πολύ τροφή για συζήτηση. Θα σας ε, δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, θα μιλήσω για εθνικές εμπειρίες, τι συμβαίνει δηλαδή στη Γερμανία. Θα σας μιλήσω επίσης και για κάποιους στόχους ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κριτική προσέγγιση για τη διαδικασία τη Μπολόνια. Διότι υπάρχει ένα χάζο μεταξύ αφενό των στόχων τη διαδικασία Μπολόνια και ε, των επιτευγμάτων τη αφετέρου. Η καθημερινή ε, προσπάθεια που γίνεται. Θέλουμε φυσικά και εμεί να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Προ το παρόν όμω βλέπουμε κάποιε πολύ αρνητικέ εξελίξει σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε ότι τα πανεπιστήμια γίνονται όλο και περισσότερο ελίτ ή γίνονται κερδοσκοπικοί οργανισμοί όλο και περισσότερο ξεχνώντα ε, τον πρωταρχικό του ρόλο που είναι η παροχή εκπαίδευση. Αυτό ε, επίση που βλέπουμε στη Γερμανία είναι ότι πολλοί κατηγορούν τη διαδικασία της Μπολόνια για τα πάντα. Ακόμη και για θέματα τα οποία προϋπήρχαν της διαδικασίας της Μπολόνια στα γερμανικά πανεπιστήμια. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τις ε, διάφορες δομές, οι είναι αρμόδιες για τον καθορισμό του νέου πανεπιστημιακού τοπίου. Πρώτα απ' όλα οι χώρες, οι χώρες οι οποίες έχουν προσυπογράψει τη Συμφωνία της Μπολόνια, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, τα Λέντρ, τα κρατήδια δηλαδή που είναι αρμόδια, αλλά και τα ε, ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι διάφορες σχολές. Έχετε λοιπόν την κατανομή των αρμοδιοτήτων και εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι βλέπουμε ότι ο ένας περτάει τον παλάκι στον άλλο σε ό,τι αφορά τις ευθύνε, Βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα γιατί δεν κινείται κανείς. Άρα, δυσαρέσκεια από την πλευρά των φοιτητών και συγκεκριμένα πέρυσι το φθινόπωρο είδαμε στις ευρωπαϊκές χώρες ότι εξεγέρθηκαν οι φοιτητέ κατά του προβλήματος αυτού και βγήκαν στους δρόμους. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, κινητικότητα, που ο σημαντικός στόχος είναι και οριζόντια και κάθετη κινητικότητα να αυξηθεί. Είναι ένας στόχος που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα και αυτό συνιστά πρόβλημα, διότι πολλές φορές η κινητικότητα περιορίζεται ε, στο εσωτερικό μιας σχολής. Ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια δεν μπορεί να περάσει από ένα κύκλο σπουδών σε έναν άλλο. Παρότι υπάρχουν κοινά μαθήματα, ε, δεν αναγνωρίζονται οι γνώσεις που έχει αποκτήσει κανείς ε, κάνοντας μια συγκεκριμένη σχολή. Παρότι μπορεί να εν μέρη να επικαλύπτεται με τα μαθήματα μιας άλλης σχολής. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια διαδικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα σας πω τι συμβαίνει στην Ομοσπονδιακή ε, Γερμανοί Θα μπορούσαν να υιοθετηθούν κάποια προπαρασκευαστικά ε, μέτρα. Δεν υπάρχει ε, μόνο το θέμα του χρόνου σε ό,τι αφορά τα προγράμματα εκμάθησης ε, γλωσσών. βέβαια, ο χρόνος είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Στα κρατήδια, στα 16 κρατήδια, υπάρχουν διαφορετικές δομές για να, για να εφαρμοστεί λοιπόν η διαδικασία της Μπολόνια. Πρέπει να υπερπηδηθούν κάποια εμπόδια που έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές δομές του κάθε κρατηδίου. Θα πρέπει λοιπόν ξεκάθαρα να πούμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας και έτσι θα βελτιωθεί και θα αυξηθεί η κινητικότητα. Και, όχι, ε, και μιλάμε τώρα για μέσα στην ίδια χώρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, ε, παραδείγματος χάρη, τα μάστερ. Μπορεί να είναι το μάθημα ε, να καλύπτει δύο ή τρία εξάμεινα και δεν μπορώ να το παρακολουθήσω και στα τρία εξάμεινα. Ή επίσης το, το περιεχόμενο. Μπορεί να είναι συγκρίσιμο το περιεχόμενο, αλλά να έχει διαφορετικό όνομα το μάθημα από μια σχολή στην άλλη. Και υπάρχει ε, πρόβλημα, ε, δεν αναγνωρίζονται δηλαδή τα μαθήματα, όχι λόγω του ότι είναι διαφορετικό το περιεχόμενο, αλλά είναι διαφορετική ονομασία τους. Επίσης, οι συμβαλόμενες χώρες πρέπει να καταπολεμήσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Δυστυχώς όμως πολλοί φοιτητέ δεν μπορούν να μεταχούν στο εξωτερικό, πολύ απλά γιατί υπάρχουν πολλοί μεγάλα εμπόδια. Πρέπει να πάνε σε πολλά γραφεία, να συμπληρώσουν του κόσμου τα φυλάδια ή δεν έχουν και τη σωστή ενημέρωση πολύ απλά για το τι συμβαίνει στα διάφορα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά την ε, ομοσπονδιακή ε, δημοκρατία, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση για τους φοιτητές ανεξαρτήτως προέλευσης ή προορισμού. Και κυρίως θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα για φοιτητές με αναπηρία. Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα, η διαβίου μάθηση. Πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο επενούμε φυσικά. Δυστυχώς όμως εδώ βλέπουμε ότι και πάλι πάρα πολλά είναι τα εμπόδια. Υπάρχουν ζητήματα χρηματοδότησης που είναι αρμοδιότητα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και των μεμονωμένων κρατών μελών. Και βέβαια θα πρέπει και τα ζητήματα που αφορούν το δίκαιο εργασίας, το δικαίωμα εργασία, θα πρέπει ε, ό,τι εμπόδιο υπάρχει να αντιμετωπιστεί χρηματοδότηση ώστε να έχουν αξιοπρεπέ ε, επίπεδο διαβίωση φοιτητέ και ούτω καθεξή. Παραδείγματο χάρη, μια φοιτήτρια που ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αρχίζει να εργάζεται και είναι μια ανύπατρη μητέρα. Θέλει να κάνει μάστερ. Δυστυχώ δεν μπορεί, δεν υπάρχει λύση. Πρέπει να βρεθεί λύση. Έρχομαι στο ε, συμπέρασμα που μπορούμε να συναγάγουμε. Τα προβλήματα που σας ε, έδειξα ε, εν είδη παραδειγμάτων θα μπορούσαν να, να μεταφερθούν και στη δομή παραδείγματος χάρη της κατανομής αρμοδιοτήτων θα έπρεπε οι αρμόδιοι να ασκούν σωστά τι αρμοδιότητες και τι ευθύνε του. Η εφαρμογή τη διαδικασία τη ε, Μπολόνια δεν δείχνει μέχρι στιγμή ότι εξελίσσεται με τον ε, σωστό τρόπο. Θα πρέπει να γίνουν απαραίτητε βελτιώσει. Φυσικά αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει ούτε να καταδικάσουμε τη διαδικασία, ούτε να ενεργούμε χωρίς συντονισμό. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία, πρέπει να εξαλειφθούν τα σφάλματα και να επιτύχουμε τους στόχους μας κατά αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάιζερ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Χάουαρντ Νιούμπι. Για 10 λεπτά. Και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και το γύρο ερωταποκρίσεων. Thank um, Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή τη φάση της ακρόασης, ε, κυρίες και κύριοι, πολλά από τα σχόλια τα οποία θέλω να κάνω έχουν ήδη γίνει. Γι' αυτό θα ήθελα να επικεντρωθώ σε πολύ λίγα αλλά σημαντικά θέματα. Και ξεκινώντας θα σας μιλήσω για τη βιωσιμότητα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη μακροπρόθεσμα, διότι τα διλήμματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε παρόντος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά δεν είναι μοναδικά, δεν αποτελούν ίδιον της Ευρώπης, ε, υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αν ήθελα να τα συνοψίσω, θα έλεγα ότι προκαλούνται από τα εξή. Πρώτα απ' όλα, όλε οι κυβερνήσει και στα κρατημέλη τη Ένωση και αλλού έχουν δεχθεί την αρχή τη βασισμένη στη γνώση οικονομίας. Αυτό θα πει ότι η μελλοντική ανταγωνιστικότητα στη δική μας περίπτωση στην Ευρώπη εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει στην Ευρώπη και από αυτήν την έννοια τα πανεπιστήμια έχουν διπλή σημασία, διότι όπως ακούσαμε ήδη στον πανεπιστημιακό κόσμο ε, υπάρχει μεγάλο ποσοστό γνώσης που παράγεται και βάσει σε αυτή τη γνώση, ε, σε αυτή τη γνώση μάλλον βασίζεται και η οικονομία μας. Θα πρέπει λοιπόν τα πανεπιστήμια να παρέχουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες στους φοιτητές και να τους διδάσκουν κατά τρόπο ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ε, για την παραγωγικότητα αυτές τις γνώσεις που θα αποκτήσουν. Λόγω της σημασίας λοιπόν που έχουν τα πανεπιστήμια σε αυτή τη διάσταση ε, και στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, δεχόμενοι, δεχόμενοι αυτά τα επιχειρήματα προσπαθούν ε, να παράσχουν μαζικά, μιλάμε για τη μαζικοποίηση τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ε, των, της ανώτατης εκπαίδευσης Συγχρόνω έχουν στόχο και την αύξηση της ποιότητας τη εκπαίδευση στα πανεπιστήμια και πάλι ανά την Ευρώπη. Οι κυβερνήσει τα κράτη-μέλη θέλουν να επιτύχουν και τα δύο. Και όχι μόνο και τα δύο, αλλά και ταυτόχρονα μειώνοντας το κόστος ε, που θα βαρύνει το φορολογούμενο διότι ξέρουμε ποιε είναι οι προτεραιότητες για τις δημόσιες δαπάνες, ιδίω ε, στα πλαίσια του παρόντος ε, οικονομικού κλίματος. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο κινείται η εκπαιδευτική πολιτική, έχουμε τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και έχουν γίνει προσπάθειες επίλυσης των διαφόρων των δυσκολιών που έχουν προκύψει. Σε κάποιες χώρες πράγματι επλήγει η ποιότητα. Σε κάποιες χώρες αυτό το ποσοστό της ε, επέκτασης, διεύρυνσης της συμμετοχής των φοιτητών δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θα ήταν σε άλλες περιπτώσεις. Και σε κάποιες χώρες, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, αυτό το δίλημα επιλύθηκε μέσω της ε, αναζήτησης περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως στην ε, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που υπάρχει συνεχή συζήτηση και αιτήματα για ανώτερη εκπαίδευση και καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να αναμένει κανείς ότι θα καλύψει το πλήρες κόστος. Έχουμε λοιπόν αυτά τα διλήμματα. Αυτά θα μας συνοδεύουν τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. Δύσκολα δηλαδή για το προβλέψιμο μέλλον θα αλλάξει κάτι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο σημείο που θέλω να σχολιάσω. Στην Ευρώπη νομίζω ότι καταλαβαίνουμε με οξύμια θα έλεγα, ε, τη μεταβατική φάση που περνούν τα πανεπιστήμια από ε, το μοντέλο του Χάμπολ του 19ου αιώνα ε, στο σημερινό μοντέλο. Ο Χάμπολ πώς αντιλαμβανόταν τα πανεπιστήμια και συμπεριλαμβανόταν στην ε, συμπεριλαμβανόταν στο ρόλο του Πανεπιστήμιου η έρευνα εκτός της εκπαίδευσης αλλά επίσης ε, ε, υπήρχε ένας διαχωρισμός των πανεπιστημίων από την κοινότητα από την επιμόλυνση τους ε, με τον απλό κόσμο. Τον 20ο αιώνα είδαμε λοιπόν να είναι λίγο απερχιωμένο ορισμένα πανεπιστήμια και επειδή υπήρχε αυτό το ζήτημα της οικονομίας της γνώσης που έχει ε, αποτελέσει κομβικό πλέον θέματα πανεπιστήμια στον 21ο αιώνα πρέπει να κάνουν αυτή την προσαρμογή, αυτή τη μετάβαση που είναι επώδυνη αλλά είναι αναγκαία και συνεχίζεται, ακούσαμε και από προλαλήσαντες ακόμη και σήμερα αυτή η μετάβαση και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την αλλαγή που, έχουν, ε, που έχει επισυμβεί στα πανεπιστήμια πριν από μία γενιά, ε, κυρίαρχο ρόλο των πανεπιστημίων ήταν η διδασκαλία και η έρευνα γινόταν ε, στον ε, υπόλοιπο χρόνο, στα περιθώρια. Ό,τι έμενε δηλαδή. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, αναγνωρίζουμε ότι τα σύγχρονα πανεπιστήμια λειτουργούν πολύ πιο πολύπλοκα. Ναι, με διδασκαλία, αλλά όπω ακούσαμε θα πρέπει να μιλάμε ουσιαστικά για διαβίου μάθηση. Αναγνωρίζουμε ότι λόγω τη αλλαγή, στην κοινωνία, στην οικονομία υπάρχουν φοιτητέ που θέλουν να συνεχίσουν τι σπουδές από καιρού καιρών σε όλη τη διάρκεια τη επαγγελματική σου σταδιοδρομία, σε μερική απασχόληση κάποιε φορές, πλήρω σε πλήρη χρόνο, ε, μέσω ίσω της εξαποστάσεω μάθηση, της, ή του e-learn, της ηλεκτρονικής μάθησης. Η πολυπλοκότητα λοιπόν και η διαφοροποίηση αυξάνονται και θα συνεχιστεί αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει η εκπαιδευτική πολιτική να το λάβει υπόψη. Ναι. Δεύτερον, ακούσαμε ότι είναι πολύ σημαντική και η έρευνα και είναι ε, φυσικά αλήθεια αυτό και στην Ευρώπη και στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει και η έννοια τη μεταφορά γνώση, ώστε όλοι να μπορούν να αξιοποιούν τη γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια και να έχουν πρόσβαση σε αυτή με τον όσο τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Και βέβαια θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα και την κοινωνική ένταξη, ε, διότι είναι ένα μοχλό κοινωνική ένταξη στα πανεπιστήμια όλο και περισσότερο και όλοι όσοι αποφελούνται τις ανώτερες εκπαίδευση παρά του οικονομικού κοινωνικού υποβάθου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και για το δικό του συμφέρον και για το συμφέρον τη κοινότητα εν γέννη. Επίση, συνεισφέρουν τα πανεπιστήμια στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη και τέλο ε, συμβάλλουν στην κοινωνία των πολιτών διότι είναι όλο και πιο σημαντικά ιδρύματα ε, που είναι μεταξύ ε, του κράτου και του πολίτη και θα πρέπει να δούμε τι κάνει την ανώτερη εκπαίδευση ανώτατη ή ανώτερη είναι να μπορέσουμε να προαγάγουμε την αγωγή του πολίτη, την ανεκτικότητα, τη δημοκρατία, τον ορθολογισμό και τα λοιπά Όλε αυτέ τι αρχέ, να τι εμφυσίσουμε στου φοιτητέ. Όλα αυτά λοιπόν ο ρόλος του σύγχρονου πανεπιστημίου. Έχουμε ένα δίλημα, έχουμε ένα πρόβλημα στην Ευρώπη. Το εξή, ότι κανένα πανεπιστήμιο, κανένα πανεπιστήμιο δεν έχει επαρκεί σπόρου ώστε να επιτύχει όλου αυτού του ρόλου ταυτόχρονα. στο παγκοσμιοποιημένο επίπεδο αριστείας και όχι στο τοπικό επίπεδο αριστείας. Αυτό είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα πανεπιστήμια θα πρέπει να επιλέξουν, να επικεντρωθούν, να εντοπίσουν τι, σε τι είναι καλύτερα και εκεί να επικεντρωθούν για να είναι πιο ανταγωνιστικά ε, σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Και άλλα ε, τμήματα του πανεπιστημιακού ε, κόσμου να επικεντρωθούν σε άλλους τομείς. Τέταρτο λοιπόν σημείο. Αν θέλουμε τα πανεπιστήμια να εντοπίσουν τα ισχυρά του σημεία, να επικεντρωθούν σε αυτά, να επενδύσουν σε αυτά και να είναι βιώσιμα, θα πρέπει να είναι αυτόνομα. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις επιλογές. Και βέβαια η αυτονομία θα πρέπει να συνοδεύεται και με την υποχρέωση λογοδοσίας. Το αναγνωρίζουμε αυτό, αλλά στην Ευρώπη, αν δει κανεί τι συμβαίνει, θα διαπιστώσει ότι σήμερα ακόμη τα πανεπιστήμια δεν είναι παρκώς αυτόνομα, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτές τις κρίσιμες επιλογές και η ανώτερη και ανώτερη εκπαίδευση στην Ευρώπη πλήττεται από αυτό. Και η απόδειξη είναι ότι εν γέννη σε όλο τον κόσμο Όσο πιο αυτόνομα είναι τα πανεπιστήμια, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο ανήκουν. Δεν ακούστηκε και πολύ όρος παγκοσμιοποίηση αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε ένα στον άλλο εδώ στην Ευρώπη ότι οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης επηρεάζουν ε, τα πανεπιστήμια με παρόμοιους τρόπους όπως επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τους, ε, τις οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα. Ανταγωνιζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο για να έχουμε, ε, αν θέλετε, το δίκαιο μερίδιο σε ταλέντα, σε ό,τι αφορά ε, τους ε, ερευνητές, ό,τι αφορά τους πανεπιστημιακούς και κυρίως ό,τι αφορά τους ταλαντούχους φοιτητές. Οι πιο ταλαντούχοι καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές είναι και οι πλέον κινητικοί. Αυτό συμβαίνει ισχύω σε μεταπτυχιακό επίπεδο και συμβαίνει όλο και περισσότερο και στο δευτεροβάθμιο εκπαίδευση. Και είναι πολύ σημαντικό, είναι ζωτική σημασία στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να έχουν το δικό τους μερίδιο, ε, ένα μεγάλο ε, μερίδιο ταλέντου και ταλαντούχων ερευνητών καθηγητών κτλ. Επίσης ε, η παγκόσμια ηθαγένεια, οι αρχές της παγκόσμιας ηθαγένειας είναι κάτι που θα πρέπει να το ενστερνιστούν οι Ευρωπαίοι φοιτητέ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, τις παγκόσμιες προκλήσεις ό,τι αφορά τη δημοσία υγεία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή και ούτω καθεξής. Και έτσι έρχομαι στο τελευταίο σχολείο μου. Ο προλαλής σας ε, μίλησε πολύ για τη διαδικασία της Μπολόνη και τις δυνατότητες που διανοίγονται και είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει στην ατζέντα της Μπολόνια να προσθέσουμε και κάποια από τα ζητήματα που ανέφερα εγώ. Και δει αυτό που σημείωσε και ο προλαλής, να εξασφαλίσουμε όπου μπορούμε ότι είναι νέοι και όχι τόσο νέοι ε, Ευρωπαίοι που μπορούν να αποφεληθούν από την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση να έχουν την ικανότητα να έχουν πρόσβαση, τη δυνατότητα μάλλον να έχουν πρόσβαση στην ανώτερη ανώτατη εκπαίδευση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση δεν θα είναι περιορισμένη ε, στο πλαίσιο ε, του σημερινού οικονομικού κλίματος. Θα πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον του Ευρωπαίου πολίτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή. Ευχαριστούμε για όλες τις εισαγωγές. Στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη όπου σπούδαζα στο τέλος της δεκαετίας του 80 από όπου βγήκαν πολλά ταλέντα και πολλές καινούργιες ιδέες Έχω μερικές σύντομες ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν από τη θέση που βρίσκονται. Ο κύριος Μπεν Πάτον πρώτος, μετά Μπερλιγκέρ, ε, Σουέρ. Θα πάρουμε τις ερωτήσεις στην αρχή, έναν κύκλο ερωτήσεων και μετά θα απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εκπρόσωπο των φοιτητών αλλά και του άλλου, γιατί έθεσαν το θέμα τη καινοτομία. Το πρόβλημα των πανεπιστημίων σήμερα σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε τα νέα στοιχεία που υπάρχουν. Μια πρώτη ερώτηση. Δεν θα έπρεπε να επενδύσουμε περισσότερο για να έχουμε πιο μεγάλη πρόσβαση για τους φοιτητές που δεν έχουν χρήματα να μην πάει χαμένη η ξυπνάδα επειδή οι κοινωνικές συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδέ. Σήμερα στην κοινωνία της γνώσης που ζούμε, αυτό δεν είναι θέμα πια μόνο ε, ισότητας και δικαιοσύνης, είναι και λειτουργικό πρόβλημα για την ίδια την κοινωνία, στο σύνολό της. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Η διαδικασία της Μπολόνια. Τη λέμε διαδικασία γιατί δεν είναι ένας νόμος που έρχεται από πάνω. Είναι μια διαδικασία bottom-up όπως λέμε, από κάτω προς τα πάνω. Αντίθετα, οι κυβερνήσεις το εφάρμοσαν top-down, από πάνω προς τα κάτω, καπελωτικά. Σε αντίθεση με την ίδια την ιδέα που λέει να πάμε προς ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Ο φοιτητή επεσήμανε τα διάφορα προβλήματα και υπάρχουν πάρα πολλά ασθενή σημεία, αλλά η διαδικασία είναι μη αντιστρέψιμη. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Και τι ακούμε, ακούμε παράπονα, γκρίνια, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα όμω δεν τα δημιουργήσει η διαδικασία τη Μπολόνια. Υπάρχουν σε ένα πανεπιστήμιο που αλλάζει και σε ένα τμήμα των σώματος των διδασκόντων που δεν θέλει να, ανάξει, να αλλάξει την διδακτική του δράση έναντι εκατομμυρίων φοιτητών. Δεν μιλάμε για δεκάδες και χιλιάδες φοιτητές. Μια βαθιά καινοτομία είναι αυτή. Μια νέα μεγάλη αλλαγή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Το χωράμε τον επόμενο συνάδελφο. Thank you for the opportunity to, to take the floor. Ευχαριστώ που μου δίνει ευκαιρία. Είμαι από τα Ευρωπαϊκά Εμπορικά Επιμελητήρια και χαίρομαι που δίνεται η δυνατότητα όπως έγινε να συμβάλλουμε στο κείμενο το οποίο συνέτρεξε ο κύριος Σμιτ. Πολλά ευχάριστα πράγματα άκουσα σήμερα από τους ομιλητές. Αυτονομία, ευελιξία, ε, να είναι υπόλογα τα πανεπιστήμια. Όλοι συμφωνούμε με τους στόχους αυτούς, αλλά το κύριο μήνυμα για μας είναι η απασχολησιμότητα. Ο καθηγητής από το Λίβερπουλ μας είπε ότι ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι να παράγει γνώσεις και ανθρώπους που μπορούν να μετατρέψουν αυτή τη γνώση, να την αξιοποιήσουν, να τη χρησιμοποιήσουν θετικά. Στην παραγωγή αυτών των ανθρώπων, με αυτές τις δεξιότητες, εμείς θεωρούμε ότι η ε, απασχολησιμότητα πρέπει να είναι το σλόγγαν, το βασικό σύνθημα, το μάντρα, όπω θα λέγαμε, των πανεπιστημίων. Αν λοιπόν εντοπίζουμε το πρόβλημα και τι χρειάζεται για βελτίωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δύο σημαντικά εμπόδια στον δρόμο αυτό. Το ένα είναι ότι το νομικό σύστημα σε μερικές χώρες δεν επιτρέπει στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις να συνεργαστούν. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να πάρουν μέρος στην διαχείριση των πανεπιστημίων σε μερικές χώρες και ακόμη πιο δύσκολο από εκπροσώπους των επιχειρήσεων να ε, επηρεάσουν κατά κάποιο τρόπο τη διδακτέα ύλη. Έχουμε PhD σε ορισμένες χώρες. όπου απαγορεύεται εντελώς ο ιδιωτικός τομέας να παρέμβει όσον αφορά τη διδακτέα ύλη. Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν, ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής, τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο γι' αυτό, αν είναι δυνατή η ευρωπαϊκή λύση. Και το δεύτερο εμπόδιο, φραγμός, είναι ότι τα πανεπιστήμια και οι πανεπιστημιακοί αξιολογούνται με βάση τα δικά τους κριτήρια. Τα δημοσιεύματα και η έρευνα, ακούσαμε, είναι το Άγιο Δισκοπότηρο των περισσότερων πανεπιστημίων. Δεν λέω, είναι και θα είναι σημαντικό, αλλά και η απασχολησιμότητα θα πρέπει να είναι κριτήριο κλειδί προκειμένου να αξιολογήσουμε ένα πανεπιστήμιο και συμφωνούμε με, αυτό που είπε ο κύριος Σμιτ πριν ότι χρειάζεται παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των ε, φοιτητών αυτών που αποφύτησαν, βρήκαν τη δουλειά που θέλανε, βρήκαν δουλειά καταρχήν και να μετρείται η επιτυχία των πανεπιστημίων με βάση και αυτό. Δεύτερη ερώτησή μου λοιπόν είναι τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να αξιολογούνται με βάση κριτήρια απασχολησιμότητας. Επίσης, χάρη, θα μπορούσε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ιεράρχηση που να, να μην στηρίζεται μόνο σε δημοσιεύματα και έρευνα, αλλά και στην σταδιοδρομία και την απασχολησιμότητα των αποφύτων των πανεπιστημίων. Και πιστεύουμε ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ σημαντικά να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα ιεράρχηση. Ευχαριστώ και πάλι που μου δώσετε την ευκαιρία να σα μιλήσω. Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σμιτ για την εξαιρετική του εισήγηση. Είναι... Ήθελα να αναφερθώ στην τελευταία παρέμβαση του κυρίου Χάουαρτ που πραγματικά με ενθουσίασε. Μας έδωσε μια εξαιρετική πανοραμική εικόνα του τι ισχύει στο χώρο των πανεπιστημίων και στην έρευνα στην Ευρώπη. Αυτό που με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερω είναι η αυτονομία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Όταν μιλάμε για αυτονομία, είναι σαν να μιλάμε λίγο για για τους φαλακρούς που έχουν ε, λίγα μαλλιά και κάποιες φορές είναι και κατσαρά. Θα πρέπει λοιπόν όταν μιλάμε για ένα πενεπιστήμια να σκεφτούμε κατά πόσον ε, υπάρχει ευθύνη έναντι των κοινωνιών και του οικονομικού συστήματος όσο πιο ανεξάρτητα είναι τα πανεπιστήμια, τόσο πιο αποτελεσματικά είναι στο ρόλο τους. Ο ο Σερ Χάουαρτ προέρχεται από την ε, Μεγάλη Βρετανία και από ένα χώρο που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος να μιλάει για τέτοια θέματα. Είδαμε ότι η διαδικασία της Μπολόνια υλοποιείται σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην κεντρική Ευρώπη ακόμα παρουσιάζουμε αρκετές καθυστερήσεις. Το πρότυπο Humboldt, που θα έπρεπε να αποτελεί ένα παράδειγμα, βλέπουμε ότι δεν επιτρέπει πάντοτε να παρακολουθήσουμε πλήρως τη διαδικασία της Μπολόνια. Υπάρχουν ακόμα πολλοί φραγμοί μερικά από τα πανεπιστήμια περιφράσονται στο χώρο της ίδιας τους της αυτονομίας. Η δημιουργία λοιπόν σχέσεων με την κοινωνία και την ε, οικονομία της αγοράς είναι ζωτικής είναι ζωτική ανάγκη. Χρειάζονται πολλές προσπάθειες λοιπόν για να απτυχθούν αυτοί οι δεσμοί και να υπάρξει και διασύνδεση με την έρευνα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό ανεξάρτητα προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και αποτελεσματικότητά τους. Όμως θα πρέπει να υπάρξει και το κατάλληλο περιβάλλον για να συμβεί αυτό. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον Σερ ε, Χάουαρτ Νιούμπι κατά πόσον οι κυβερνήσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν να ευνοήσουν τη δημιουργία αυτού του περιβάλλοντο για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου να εξυγχρονιστούν εγκαίρω στην Ευρώπη και σε σχέση με τον ανταγωνισμό με τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε. Πολύ καλή αρχή. Τώρα λοιπόν που έχουν τεθεί οι ερωτήσει, ποιο από εσά θέλει να αρχίσει. Ήταν αρκετά τα ερωτήματα, νομίζω υπάρχουν για όλους. ίσως να αρχίσουν ε, οι φοιτητέ. πρώτοι. Κύριε Κάιζερ και μετά οι καθηγητές. Και θα συνεχίσουμε μετά τη συζήτηση. Το πρώτο ήταν ε, χρήματα και για τους φτωχούς φοιτητέ. Λογικό είναι αυτό. Από τη που άνοιξαν τα πανεπιστήμια σε όλους, στους ανθρώπους, που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, το χρήμα είναι πάντα ένα λεπτό θέμα αλλά τελικά είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Πρέπει να υπάρχει μια δομή προκειμένου να γίνει αυτή η επένδυση. Θα διευκολυνθούν οι φοιτητέ στην πρόσβαση και θα βοηθηθούν και οι καθηγητές για την έρευνα. Είναι πολιτική βούληση. Είναι αξία η εκπαίδευση για τον πολιτικό ή όχι. Στη Γερμανία δεν δίνεται μεγάλη σημασία στην ε, εκπαίδευση ούτε επαρκή χρήματα. Μετά ακούσαμε για την έννοια απασχολησιμότητα. Ότι δεν λαμβάνεται πάντα υπόψη. Και θα πρέπει να υπάρχει πιο στενή σχέση με τον χώρο εργασία. Πάντως δημιουργούνται νέες θέσει ε, εργασία με τον Πανεπιστήμιο. Χθε ένας Ε, η κοινωνιολογία Φερρυπίνου δημιουργεί νέες θέσει απασχόληση, μου είπε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τα πανεπιστήμια έχουν λέγει, αλλά δεν είναι, δουλειά του δεν είναι να ζουν σε έναν χώρο που αυτοί να ρυθμίζουν, αλλά να είναι ανεξάρτητα. Αυτονομία είναι μια αμφίσιμη έννοια. Γιατί μπορεί να έχουμε ζω σε ένα κρατήδιο που έχουμε τρία πανεπιστήμια που είναι εντελώ ανεξάρτητα και σε καμία σχέση το ένα με το άλλο. Φυσικά χρειάζονται αυτονομία τα πανεπιστήμια, από την άλλη μεριά χρειάζεται όμως και συγκρισιμότητα. Η προβληματική του Πανεπιστημίου Humboldt, δηλαδή ένα πανεπιστήμιο για την ελίτ, είναι και αυτό μια τάση που υπάρχει, που μπορεί να τη δει κανεί αν θέλει κριτικά. Um, Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο ερώτημα για την ανάγκη επένδυσης, ε, για τη δυσονοϊκή πρόσβαση. Φυσικά και συμφωνώ απόλυτα σε αυτούς τους χαλεπούς οικονομικούς ε, καιρούς, εάν ε, η προτεραιότητα αν θέλουν να δαπανίσουν κάποια χρήματα οι κυβερνήσει στον τομέα τη εκπαίδευση είναι για του φοιτητέ που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και βέβαια ε, όσοι έρχονται από υπόβαθρο, από γονεί πιο εύπορου, θα μπορούσαν ίσω να πληρώσουν κάποια ποσά. Αλλά τέλο πάντων είναι λίγο επίμαχο και ε, το όλο θέμα. Σε ό,τι αφορά τον ε, κύριο από το Europe Chambers, ο οποίος μίλησε για την απασχολησιμότητα, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η Επιτροπή, η Κομισιόν, δρομολόγησε ένα πιλωτικό σχέδιο Multirank για την κατάταξη των Ευρωπαίων επενδύσεων και ήμουν ε, σύμβουλος. Η απασχολησιμότητα είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν. Είναι Πολύ τεχνικό και πολύπλοκο θέμα βέβαια και ίσως χρειαστεί πολλή χρόνο μέχρι ότου γίνει αυτή η κατάταξη και ίσως να μην είναι και μία ενιαία κατάταξη. Η απασχολησιμότητα πάντως λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και μπορώ να σας αναφέρω επίσης ότι η Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων σκοπεύει να κάνει και μια κατάταξη των κυβερνήσεων σε σχέση με την αυτονομία που δίνουν στα πανεπιστήμια της χώρας τους. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της αυτονομίας. Ε, ερχόμαι στην τρίτη παρέμβαση. Φυσικά και δεν είναι αυτός σκοπός η αυτονομία. Φυσικά και δεν πρέπει να είμαστε εξω, εκτός κοινωνίας. Έχουμε ευθύνε και προς την οικονομία και προς την κοινωνία. Όπως σας είπα απλά, ο στόχος είναι να μπορούν να επιλέγουν τα πανεπιστήμια, να μπορούν να βρουν το δικό τους ρόλο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση τα ισχυρά του σημεία. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλα ε, στον ίδιο βαθμό τα πανεπιστήμια. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούν τα ισχυρά του σημεία και για να το κάνουν αυτό, κατά την άποψή μου, θέλουν στα περισσότερα κράτη-μέλη περισσότερη και όχι λιγότερη αυτονομία. Κύριε Γκάμπριελ, θέλετε το λόγο. Μία ακόμη παρατήρηση σχετικά είναι ότι ένα γενικό πρόβλημα των ε, πανεπιστημίων και σε σχέση τους με τις επιχειρήσεις είναι ότι συνεχώς υπάρχουν προτάσεις για κάποιες προσθήκες, νέες ιδέες για τους κύκλους μαθημάτων. Ο στόχος είναι να υπάρξει ανταλλαγή και ενίσχυση της ε, μετάδοσης δεξιοτήτων και των ε, γνώσεων των πρακτικών. Αυτό το δίλημα λοιπόν, το, το ποια επιλογή θα προκρίνουμε, δεν έχει επιληθεί ακόμη. Τι θεωρούν ε, τα πανεπιστήμια ως ε, δεξιότητες που μπορεί να μεταφερθούν. Σίγουρα υπάρχει ένταση μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των διαφορών χωρών. Διαφορετική αναγνώριση των πτυχίων και των διπλωμάτων. Όλο αυτό δυσχεραίνει το την ε, αρμονική συνεργασία. Ευχαριστούμε. Θα έχουμε τώρα τρεις παρεμέροντες πάλι. Ε, Κύριε Σφέρ, θέλετε να επανέλθετε. Δεν θα σας ικανοποιήσει η απάντηση. Θέλετε να θέσετε πάλι την ερώτησή σας, γιατί δεν φαίνεται να λάβετε την απάντηση που θέλατε. Πολύ σύντομα. Να σχολιάσω την απάντηση. Μπορώ. Ευχαριστούμε. Όπως και εσείς είπατε, τα πανεπιστήμια σίγουρα χρειάζονται αυτονομία. Όμως τον 21ο αιώνα τα πανεπιστήμια θα αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο ευθύνε σε σχέση με την αποστολή τους. Δεν έχουν πια το μονοπόλιο στην αγορά, ούτε στην κατοχή της γνώσης. Η οικονομία δεν ανατρέχει πλέον μόνο στα πανεπιστήμια για να λάβει αυτά που χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα μάλιστα και να τους συγχαρώ γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι παρουσιάσεις. μας βοήθησαν να δούμε διαφορετικές οπτικές γωνίες ό,τι αφορά και τα αποτελέσματα της διαδικασίας της Μπολόνιας αλλά και σε ό,τι αφορά τη σημασία της στρατηγικής Λισαβόνας. Αναφέρθηκε ο ρόλος των πανεπιστημίων για την επίτευξη των στόχων που έχει ορίσει η στρατηγική της Λισαβόνας. Και νομίζω ότι στον τομέα αυτό σημασία δεν έχει μόνο κοινωνική συνοχή. Σημασία έχει επίσης ε, και η καλύτερη ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνα στην Ευρώπη, γιατί στη στρατηγική της Λισαβόνας υπάρχει αυτός ο στόχος. Ε, τα πανεπιστήμια λοιπόν είναι υπεύθυνα και πρέπει να επιτελέσουν ε, το ρόλο τους για την επιτευξή αυτού του στόχου. Στην παρουσίαση που ακούσαμε από την κυρία από τη Ρουμανία διαπίστωσα ότι έκανε μια πολύ σωστή ανάλυση του ρόλου και τις σχέσεις που θα πρέπει να έχουν τα πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις. με στόχο εναρμόνιση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να ρωτήσω την κυρία Κάρπ που έχει και πολύ καλή εμπειρία στο θέμα ως ερευνήτρια στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και ως καθηγήτρια πανεπιστημίου. Θέλω λοιπόν να τη ρωτήσω. Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο παράγοντας που καθορίζει τον πολύ διαφορετικό βαθμό ε, κατά τον οποίο οι φοιτητέ όταν πάρουν το δίπλωμά τους ε, ανταποκρίνονται στις, ε, ή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσει τη αγορά. Να απαντήσω τώρα. Ευχαριστώ Ευχαριστώ τον κύριο Κάιζερ που εστίασε και πάλι τη συζήτηση στην διαδικασία της Μπολόνια διότι θεωρώ ότι όντω όταν μιλάμε για το μέλλον των πανεπιστημίων και τις προκλήσεις πρέπει να αναλύσουμε τι έγινε με την διαδικασία Μπολόνια μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στους στόχους. Επετεύχθησαν όμως και αυτό που προσπάθησε να καταστήσει σαφές ο κύριος Κάιζερ είναι ότι στο δρόμο αυτό τη εφαρμογή αυτή τη διαδικασία των στόχων τη Μπολόνια δεν έχουμε προχωρήσει πολύ όσο θα θέλαμε. Για να μην πω ότι το τρένο μπορεί να κινείται και σε λάθο κατεύθυνση. Επιγόντω λοιπόν ω Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να φροντίσουμε, με τι λίγε βέβαια αρμοδιότητε που έχουμε για το θέμα αυτό, να φροντίσουμε το πώ να πετύχουμε τους στόχους της Μπολόνια και ταυτόχρονα οι σπουδές να είναι ανοιχτέ για τους φοιτητές και τις φοιτήτρες και για την κοινωνία. Όλοι να κερδίζουν. Ο καθηγητής Νιούμπαρ είχε δίκιο για την κοινωνική την κοινωνική ευθύνη των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια συμβάλλουν στην κατάρτιση στην εκπαίδευση, στη δημιουργία μιας κοινωνίας πολιτών. Δεν είναι μόνο τους τα πανεπιστήμια στον κόσμο, μόνο για να δίνουν επιστημονικές γνώσεις. Έχουν κοινωνική ευθύνη επίσης. Και η διδαχή είναι ένα κομμάτι αυτής της κοινωνικής ευθύνης. Και θέματα ηθικής θα πρέπει να συναπαντούν και τα πανεπιστήμια και με τους φοιτητές. Βέβαια το πρόβλημα είναι όπως γίνεται σε πολλές χώρες η μετάφραση της μεταγραφή της διαδικασίας της Μπολόνια δημιούργησε ένα κορσέ που δυσκολεύει τις σπουδέ. Δεν μπορεί κανείς να κοιτάξει ούτε αριστερά ούτε δεξιά όσον αφορά την ειδικότητα που έχει επιλέξει. Αν περιοριζόμαστε έτσι στενά, ε, τότε ακριβώς η κοινωνική ευθύνη που θα έπρεπε να δώσουν και να έχουν στα μάτια τους μπροστά τα πανεπιστήμια, τη χάνουμε λίγο. Γι' αυτό η ερώτησή μου και πάλι προς όλους, τι δυνατότητα βλέπετε μια επανακατεύθυνση του συστήματος, της διαδικασίας αυτής, έτσι ώστε την ευθύνη αυτή έναντι μιας κοινωνίας των πολιτών εκ μέρους των πανεπιστημίων να ενισχυθεί προκειμένου να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσω την πρόεδρό μας που επανήλθε, την κυρία Πακ. Τρεις είναι ακόμη οι ομιλητές. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ όλους τους εισηγητές. Θα έλεγα ότι συμφωνώ πάρα πολύ με τα όσα είπε ο κύριος Βέρ και μετά όσα είπε εκπρόσωπο του Euro Chambers. Νομίζω ότι αυτή την εποχή δεν είναι σε 100% στην κοινωνική πραγματικότητα οι κοινωνίε της Ευρώπης και μιλώ κυρίω για τα ισπανικά πανεπιστήμια, ίσω για τα πανεπιστήμια του Νότου τη Ευρώπη που γνωρίζω ω περιοχή. Υπάρχουν ορισμένα πραγματικά προβλήματα για να έχουμε αυτή την πραγματική κινητικότητα μεταξύ του κόσμου των πανεπιστημίων και του κόσμου των επιχειρήσεων. Υπάρχουν ζητήματα νομικά κτλ. Υπάρχουν και ζητήματα ε, πρόσληψη ε, πανεπιστημιακών υπάρχουν ε, ε, διάφορες διαδικασίες για να πάρει κανείς ε, τη θέση του καθηγητή. Θα έλεγα ενδογαμικές διαδικασίες, δηλαδή υπάρχουν σχέσεις φιλίας και όχι τόσο αξιοκρατικά κριτήρια τα οποία καθορίζουν το ποιος θα λάβει το, τη θέση του καθηγητή στο πανεπιστήμιο ως επιχειρηματίας και δικηγόρος πρώτο ασχοληθώ με την πολιτική. Θεωρώ πολύ δύσκολο ένας φοιτητής ο οποίος βγαίνει από το πανεπιστήμιο να είναι πραγματικά προετοιμασμένος ε, για να φέρει σε πέρας ε, τα καθήκοντα που θα έπρεπε να μπορεί να φέρει σε πέρας. Ένας εξαιρετικός φοιτητής για μένα δεν είναι αυτός ο οποίος έχει πολύ υψηλές θετικές θεωρητικές γνώσεις, αλλά αυτός που έχει γνώσεις που θα το επιτρέψουν να είναι χρήσιμος για την κοινωνία και βέβαια θα μπορεί να κερδίζει το ψωμί του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι η κοινωνία θα πρέπει γενικά να προσαρμόζεται όλο και δυνατόν, ε, όσο το δυνατόν περισσότερο προ αυτή ακριβώς την προετοιμασία. Φυσικά και έχουν ευθύνη τα πανεπιστήμια, αλλά και οι ε, εταιρείε και δι δημόσιε εταιρείε που κοστίζουν και πολλά χρήματα στο φορολογούμενο θα έπρεπε να έχουν ένα ρόλο, αλλά και η κοινωνία γενικώ θα έπρεπε να είχε λόγο σε ό,τι αφορά τη διδακτία ύλη των πανεπιστημίων, την κατάρτιση, την κινητικότητα των καθηγητών, τον βαθμό προετοιμασία ε, και ετοιμότητα των φοιτητών και το καθεξής. Θα σα δώσω ένα μικρό παράδειγμα που δεν έχει καμία σχέση με τι επιχειρήσει. Ένα φίλο μου καθηγητή Λατινικών στο Πανεπιστήμιο τη Βαρκελόνη μου έλεγε ότι εμεί όταν σπουδάζαμε όταν τελειώναμε το σχολείο, ξέραμε πολύ περισσότερα λατινικά από ό,τι ξέρουν οι φοιτητέ ε, ε, που σπουδάζουν λατινικά στο πανεπιστήμιο. Το επίπεδο λοιπόν διδασκαλία στα πανεπιστήμια δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαιρετικό και σε καμία περίπτωση δεν είναι προσαρμοσμένο στι πραγματικότητε, τι κοινωνικέ. Θα ήθελα αν οι ειδικοί εμπειρογνώμονε μα θα μπορούσαν να μα κάνουν συγκεκριμένε προτάσει. Η θεωρία είναι πολύ καλή, πολύ ωραία μα τα εξήγησαν, αλλά τι μπορούν να κάνουν τα πανεπιστήμια για να προσαρμοστούν ε, σε αυτέ τι κοινωνικέ πραγματικότητε και στι ανάγκε τη κοινωνία. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σμιτ και την κυρία Μαδουρέλ για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε σήμερα. Στο Κοινοβούλιο, σε πολλές επιτροπές, συζητούμε τα ίδια ακριβώς ε, θέματα. Και εγώ προσωπικά συνέταξα μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη χωρίς την έρευνα, την εκπαίδευση δεν έχει μέλλον. Ε, πόσο μάλλον χωρίς μια ολιστική προσέγγιση για αυτά τα ζητήματα. Θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε να μάθουμε κάτι έστω και εκ των υστέρων από, τις αμερικανικές, από την παράδοση των Αμερικανικών πανεπιστημίων που κάποιες φορές ε, επικρίναμε ότι είναι πάρα πολύ χαλαρά τα πανεπιστήμια, πάρα πολύ ανομιγένη κτλ. Όλοι είμαστε υπέρ της αμοιβαιότητας, ε, δυναμισμός, ε, ευελιξία, ελαστικότητα των πανεπιστημίων, διεπιστημονικές πτυχές κτλ. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον ε, την παρουσίαση του κυρίου Γκάμπριελ από το Πανεπιστήμιο του ΠΕΤΣ της Ουγγαρίας στην Ανατολική Ευρώπη πριν από χίλια χρόνια. Ήδη είχαν σχέσεις το ΠΕΤΣ και η Κωνσταντινούπολη. Τα πανεπιστήμια δηλαδή. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να έχουμε σήμερα στην Ευρώπη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων. Γιατί οι Αμερικανοί μπορούν πιο εύκολα να μετατρέπουν τη θεωρία σε πράξη, ε, την ιδέα σε ένα προϊόν. Γιατί εμείς στερούμε, γιατί υπολοιπόμαστε. Ε, στη Φινλανδία ίσως εμείς να είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτή τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών και αυτή την περίοδο προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε και τη διοίκηση των πανεπιστημίων. Υπάρχουν μάλιστα στη διαδικασία αυτή και κάποιοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων οι οποίοι συμμετέχουν, αλλά κάποιοι κατηγορούν ε, τη διαδικασία αυτή. Παλιά λέγανε ότι οι πανεπιστημιακοί τα ρυθμίζουν όλα. Τώρα λένε το αντίθετο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πολλές μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές, διεθνείς εταιρείες Ε, πρέπει να έχουν και αν θέλετε κάποια ανθρωπιστική ε, προσέγγιση στα διοικητικά συμβούλια, δηλαδή να μην έχουν μόνο επιχειρηματίες, να έχουν κάποιους μέχρι και θεολόγους, ε, κάποιους από άλλες δηλαδή, άλλους τομείς του επιστητού. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου και δεν ήθελα να μιλήσω γιατί σχέση με τα προβλήματα του Πανεπιστημίου βρίσκομαι σε πλήρη απογοήτευση, γι' αυτό δεν ήθελα. Πολλοί συνάδελφοι πανεπιστημιακοί που στην Ιταλία είναι βουλευτέ, ο συνάδελφο Μπερτιγκόρη υπήρξε και υπουργό, δεν θέλουν να μιλήσουν για το πανεπιστήμιο γιατί δεν ξέρουν τι να πούμε. Σα εξηγώ δηλαδή ότι υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ εθνικέ εμπειρίε ανάλογα με την πρέλευση του καθενός. Και γι' αυτό και οι απόψεις μας διαφέρουν. Πρέπει για τη σχέση επιχειρήσεις πανεπιστημίου έχω μερικές επιφυλάξεις σχετικά με το αμερικάνικο μοντέλο. Τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα να πω τώρα είναι στην έκθεση που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο είναι δυνατόν να επισημαίνονται ορισμένα σημεία που δεν είναι μόνο ιταλικά προβλήματα, νομίζω αφορούν και τις άλλες χώρες. Δηλαδή, η τάση των κυβερνήσεων να περικόπτουν τον προϋπολογισμό της παιδείας και της έρευνας. Η Ευρώπη μήπως θα μπορούσε να επιβάλλει στις κυβερνήσεις της Ένωσης την υποχρέωση τήρηση ορισμένων κριτηρίων ποσοστού του προπολογισμού για την παιδεία και την έρευνα. Γιατί αυτό που γίνεται στην Ιταλία σήμερα δεν είναι αυτό ακριβώς. Και πιστεύω παρόμοια συμβαίνουν και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ορισμένες κυβερνήσεις περικόπτουν τον προπολογισμό εκεί ακριβώς που έπρεπε να τον αυξάνουν. να το θυμίζουμε αυτό και να το θυμίσουμε στην έκθεση που θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο. Δεύτερο. Υπάρχει τάση στην Ευρώπη υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι των δημοσίων. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ίσως υλοποιούν καλύτερα τη σχέση με τις επιχειρήσεις γιατί συχνά είναι προσανατολισμένα προς την άμεση ε, εφαρμογή, α το πούμε, της τεχνολογίας. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα δημόσια πανεπιστήμια κάνουν τη βασική έρευνα, που συχνά δεν ενδιαφέρει άμεσα τη βιομηχανία. Γιατί μια πολύ βασική έρευνα, στη φυσική, στη χημεία κλπ, δεν αποδίδει κέρδη στις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και την παραμελούν. Νομίζω εμείς στην έκθεσή μας πρέπει να το λέμε αυτό και να καλέσουμε τις κυβερνήσεις να σεβαστούν κριτήρια όταν δίνουν κονδύλια στα πανεπιστήμια και στην έρευνα. Είναι επίκειται αυτός ο κίνδυνος και στην Ιταλία αλλά πιστεύω ότι και στις άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βάτιμο. Όντως πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση και την έρευνα. Τουλάχιστον όχι λιγότερα, λέει ο κύριο Βάτμα. Όχι, περισσότερα, περισσότερα, λέει η πρόεδρο. Η κυρία Μπάντι μας παρουσίασε την έκθεση της χθες για το θέμα αυτό. Δηλαδή, στη Λισαβόνα τι υπάρχει για την έρευνα, για την εκπαίδευση, την παιδεία κλπ και είδαμε ότι σε μερικέ χώρε υπάρχουν πίσω γυρίσματα, όπω σωστά επισήμανε για την Ιταλία ο κύριο Βάτμα. Η κυρία Χάνιμπαλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές για ένα πολύ διαφωτιστικό απόγευμα. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι όχι βέβαια σύγκρουση, ίσω αντιπαράθεση, αλλά κάποια ένταση μεταξύ των δύο πραγμάτων που θεωρούμε ότι κροσοπούν τα πανεπιστήμια. Το πρώτο είναι να δώσουν τα, στους φοιτητές τους τα δεξιότητες είναι απασχολήσιμη και δεύτερον η γνώση αυτή καθεαυτή και η έρευνα. Αυτά νομίζω ότι είναι τα δύο πράγματα στα οποία καταλήξαμε και ίσως πάντοτε θα υπάρχει μια ένταση μεταξύ αυτών των δύο και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να προσπαθούν να αποφασίσουν προς ποια κατεύθυνση θα απορρευθούν. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι που είπε ο καθηγητής Νιούμπι, ότι κάθε ίδρυμα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό που τα καταφέρνει καλύτερα και έτσι ίσως ε, πράγματι θα μπορέσει να κάνει καλύτερα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Και νομίζω ότι το κλειδί, και αυτό ακούστηκε επίση, είναι ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν αυτόνομα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασικό και πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της συζήτηση. αυτόματα ιδρύματα που θα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο. Εγώ ε, τη διαδικασία της Μπολόνια τη βλέπω και αυτή ως ένα πλαίσιο και θεωρώ ότι λειτουργεί και καλά. Ξέρω ότι βασίζεται στο Βρετανικό σύστημα, αλλά πράγματι ξέρετε ε, αποδίδει. Έχουμε πτυχία ε, που τα παίρνει μετά από τρία χρόνια σπουδών και είναι πολύ, πολύ καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούν περισσότερο τα πανεπιστήμια είναι τι έχει να προσφέρει με μονομένα το καθένα από αυτά. Ίσως κάποια τα καταφέρουν καλύτερα στην επιστήμη για να οδηγήσουν στην απασχολησιμότητα, κάποια άλλα μπορεί να βασίζονται περισσότερο στη γνώση και στην έρευνα. Νομίζω ότι δεν το έχουν φτάσει το επίπεδο αυτό ακόμη τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, ίσως να μην έχουν ακόμη την ικανότητα να το κάνουν. Ε, βέβαια, αυτά πρόσφατα ε, τα επεξεργαζόμαστε ε, και παρότι έχουμε από το 1200 την, την, όλη συζήτηση, ουσιαστικά και τα πανεπιστήμια. Ελπίζω κάπως να βρεθεί ο σωστός δρόμος προς τα εμπρός. Θέλω να έρθω σε κάτι ίσως βαρετό, ε, που το ακούμε πολλές φορές, γλώσσες δηλαδή. Ωραία, όλα καλά, να έχουμε το ευρωπαϊκό σύστημα, να έχουμε εναρμόνιση, μιλάμε για κινητικότητα, κινητικότητα φοιτητών, κινητικότητα καθηγητών. Η κινητικότητα όμως δεν θα αποδώσει αν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Ταυτόχρονα λοιπόν, μαζί με όλα αυτά τα οποία κάνουμε ε, στο ενώτερο επίπεδο αν θέλετε, νομίζω ότι και στα κράτη-μέλη αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να δούμε πώς μπορούμε σε αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο να δώσουμε τις γλωσσικές δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να τα καταφέρουν, να μπορέσουν να μελετήσουν σε άλλα μέρη του κόσμου, της Ευρώπης. <laughs> You are British. Και τώρα η κυρία Χάλιουελ. Ναι, γνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να μάθουμε γλώσσες και κάνουμε ό,τι μπορούμε να το πείτε στους, στους εκλογείς σας, στους υπηκόους του στέματος. Αυτές ήταν οι τελευταίες ερωτήσεις. Θα ρωτήσω από τους, θα ρωτήσω από τους ομιλητές μας να απαντήσουν, ε, αν θέλουν. Για τη διαδικασία της Μπολόνια έχει γίνει πολλή λόγος. Εγώ ήδη έχω συντάξει έκθεση σχετικά. Και οι Γερμανοί εδώ έχουν μια πολύ ισχυρή παράδοση. Ξέρετε ότι η διαδικασία αυτή μας αφορά ιδιαίτερως. Να δώσω ένα παράδειγμα. Πήγα μια φορά στη Στοκχόλμη και ένας καθηγητής πανεπιστημίου εκεί σε ένα από τα πανεπιστήμια που επισκεφτήκαμε μου είπε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη διαδικασία της Μπολόνια. Είμαστε απόλυτα προσαρμοσμένοι. Εγώ πραγματικά έμεινα άναυδη. Εντυπωσιάστηκα. Φαίνονται ότι υπάρχουν και σοβαροί λόγοι γι' αυτό. Ε, μου έδειξε μάλιστα ο καθηγητή αυτός να τι κάναμε πριν την Πολόνια και τι κάνουμε τώρα. Τα πράγματα λοιπόν δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Απλώ έχει δοθεί διαφορετικό τίτλο στα πτυχία. Στο bachelor, το πρώτο πτυχίο, το master, το μεταπτυχιακό δηλαδή και ούτω καθεξής. Με ένα πρώτο πτυχίο λοιπόν, ήδη στη Σουηδία μπορεί κανεί να αναζητήσει εργασία. Είναι πολύ χρήσιμο στι επιχειρήσει, αλλά στη Γερμανία τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έχουμε περισσότερα προβλήματα από ότι ίσω οι Βρετανοί ή οι Γάλλοι. Σω να έχουμε αντιγράψει εμεί εσά κατά λανθασμένο τρόπο, ίσω να έπρεπε να έχει γίνει το ανάποδο. Σε κάθε περίπτωση να δώσω εδώ το λόγο στον κύριο Νιούμπι, στον Σερ Νιούμπι, για να μα απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση για σήμερα. Μπορώ καταρχά να ευχαριστήσω όλου του βουλευτέ για τα γενικά του σχόλια. Νομίζω ότι μιλώ εκ μέρου όλων των συναδέλφων και ήθελα και να σα ευχαριστήσω για τη σοβαρότητα με την οποία καλύψατε το θέμα αυτό και μα ακούσατε. Διότι εδώ υπάρχουν σοβαρέ προκλήσει, δεν υπάρχουν απλέ απαντήσει, όλοι τα γνωρίζουμε και νομίζω ότι αυτό το υψηλό επίπεδο διάλογο τον θέλουμε στην Ευρώπη, πρέπει να τον συνεχίσουμε. Πολύ σύντομα Ίσως η προοπτική μου να είναι βρετανική και ιδιότυπη, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει έλλειψη πρόοδου στη διαδικασία της Βολόνια. Νομίζω ότι μάλλον καλά τα πάει η διαδικασία αυτή. Ήδη νομίζω ότι πολλά κράτη-μέλη το χρησιμοποίησαν αυτό το σύστημα ως ε, πρόσχημα για να μεταρρυθμίσουν τα πανεπιστημιακά τους ε, συστήματα. Όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ευρώπη δεν μπορούν να δράσουν ε, αυτόνομα στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα κάτι μελη και οι τοπικοί φορείς συνήθως αναλαμβάνουν το βασικό ρόλο. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έρχεται να διδραματίσει ενεργότερη συμμετοχή και οι τομεί δραστηριότητα όπου θα μπορούσε να παρεκταθεί και να καλύψει η διαδικασία τη Μπολόνια, όπω τη δίκαιη πρόσβαση, είναι τομεί που μα ενδιαφέρουν και για το μέλλον, όπω το αναφέρατε κι εσεί και συμφωνώ κατά πολύ μαζί σα. Πολύ σύντομα. η μεταφορά της θεωρητικής γνώσης ε, και η λήψη υπόψη της, ε, των αναγκών της κοινωνίας. Εδώ να μην ξεχνάμε ότι το ε, πανεπιστημιακό σύστημα ανά την Ευρώπη είναι πολύ ετερογενέ. Δεν μπορεί ένα πανεπιστήμιο να τα κάνει όλα, ούτε και θα όφιλε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει περιθώριο τα πανεπιστήμια να επιτελέσουν το έργο που κάνουν καλύτερα. Εδώ νομίζω ότι ένα δίκτυο πανεπιστημίων ε, έρχεται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Να μπορούν οι φοιτητέ στην Ευρώπη, εφόσον τα πανεπιστήμια είναι διαδικτυωμένα μεταξύ του, να μπορούν οι φοιτητέ να κάνουν ελεύθερα τι επιλογέ του. Νομίζω ότι τότε πραγματικά θα βοηθήσουμε τι μελλοντικέ γενιέ. Και όπω είπε και ο Βρετανό συνάδελφο, υπάρχει όντω ένταση μεταξύ των διαφορετικών στόχων ε, τη ανώτατη εκπαίδευση. Βεβαίω, τα πανεπιστήμια θέλουν ε, να δώσουν πτυχιούχους ε, που θα είναι ικανοί να αναλάβουν τα ενία των πανεπιστημίων από το να μείνουν άνεργοι. Αλλά η συζήτηση περί πανεπιστημίων τα τελευταία 20 χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται λίγο χρησιμοθυρική και να την αντιμετωπίζουμε μόνο από τη σκοπιά των σκοπιμοτήτων τα πανεπιστήμια, μην ξεχνάμε ότι είναι και τα θεμέλια των ευρωπαϊκών αξιών μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Δεν τρέπομαι να πω ότι πιστεύω στο ότι η αύξηση της γνώσης βοηθά και την κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Τα πανεπιστήμια υπάρχουν και για αυτό το σκοπό. Έχουμε εκπαίδευση, έρευνα, μια αντίθεση Ακριβώς από την ένταση αυτή όμως ζουν τα πανεπιστήμια. Υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον. Είναι γνωστό ότι οι καθηγητές ζουν και από την έρευνα, αλλά ζουν και από το feedback που έχουν με τους φοιτητέ. Τώρα για να έρθω σε μια ερώτηση για την κοινωνική ευθύνη που θα έπρεπε να επιτρέψει η φοιτηση στο Πανεπιστήμιο. Το πιο σημαντικό είναι το workloads, Ο μέσο οικονομολόγο στην Αγγλία δουλεύει 49,8 ώρε τη βδομάδα. Δεν μένει ο χρόνος, ούτε και κίνητρα αρκετά, προκειμένου να πάρει ενεργότερο μέρος της κοινωνία. Έπειτα, το πλαίσιο είναι πολύ στενό χρονικό περιθώριο προκειμένου να αποκτηθεί το πτυχίο. Ε, αναφέρθηκε ότι η διαδικασία της Βολόνια εξαρτάται κάθε φορά από το Ομοσπονδιακό Κρατήριο γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα ε, εξαρτάται πόσο κοντά είναι στη δομή που προτείνει η διαδικασία της Βολόνια. Μπορούμε να διδαχθούμε το ένα κράτος από το άλλο, να εφαρμόσουμε τις άριστες μεθόδους που έχουν εφαρμόσει οι άλλοι. Έχουμε πετύχει κάποια πράγματα με τη διαδικασία Μπολόνια, αλλά όντω χρειάζεται να δοθεί και μια νέα κατεύθυνση μερικέ φορέ ο κύριο Κάιζερ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κάιζερ, ο, ο επόμενο καθηγητή. Θα αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία, γιατί έγιναν πάρα πολλέ ερωτήσει, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Συμφωνήσαμε μεταξύ μα τι θα απαντήσει ο καθένα. Υπήρξε ένα ερώτημα. Περισσότερα κονδύλια για την έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση από ό,τι στο παρελθόν. Τα νούμερα στην Ουγγαρία είναι πολύ χαμηλά, 1%. Για το καθένα, πολύ μικρό το νούμερο κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω τι είναι το νούμερο στην Ιταλία ή στις άλλες χώρες. Δεν αρκούν τα χρήματα αυτά. Και μετά έχουμε ένα άλλο ερώτημα. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από τους Αμερικάνους. Κατά τη γνώμη μου, ένα δίδαγμα από την Αμερική είναι ότι η χρηματοδότηση του 1% δεν αρκεί. Οι ερευνητές κάνουν έρευνα, οι διδάσκοντες φυσικά συμμετέχουν στις τάξεις, διδάσκουν. Ένα πράγμα κάνει ο καθένας. Υπάρχει διαχωρισμός στα επαγγέλματα. Μερικοί διδάσκουν περισσότερο, μερικοί αποκλειστικά κάνουν μόνο έρευνα. Γι' αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο το αμερικανικό δυναμικό από το ευρωπαϊκό. Τέλος, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εξετάται από το θέμα και από εκεί θα επακολουθήσει η κρατική χρηματοδότηση. Όταν είναι πιο κοντά στις επιχειρήσεις, τότε οι φοιτητές θα προτιμάνε μερικές φορές. Δεν ξέρω να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια για την ιατρική, χημεία κλπ. Χρειάζεται βαρύ εξοπλισμός προκειμένου να γίνει σωστά η εκπαίδευση. Και δεν ξέρω κανένα ιδιωτικό ανάτο του Ίδρυμα που θα το ενδιαφέρε αυτού του είδου η ειδικότητα. Η κυρία Καπ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα και εγώ να δώσω κάποιες απαντήσεις σε όσα σχολιάστηκα για τα κριτήρια αξιολόγησης των καθηγητών και το κατά πόσο αυτά βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην ερευνητική τους ε, απόδοση. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Τα κριτήρια πρέπει να τροποποιηθούν για να λαμβάνουν υπόψη και την προσωπικότητα των ε, καθηγητών σε αυτή τη φάση στη Ρουμανία είμαστε στην... Ε, επεξεργαζόμαστε τη μεταρρύθμιση των διαφόρων κριτηρίων. Η αξιολόγηση στα πανεπιστήμια σαφώ δεν μπορεί να είναι απόλυτη και αντικειμενική. όμως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που διαχειρίζονται δημόσια κονδύλια θα πρέπει να υπόκειται στου ίδιου νόμου όπω άλλα ιδρύματα που λαμβάνουν κρατικής διδότησης. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μην είναι τα κριτήρια αυτά απόλυτα, ιδίω ω προ τι οικονομικέ ανάγκε και τον οικονομικό τομέα. Τώρα, γιατί υπάρχουν τέτοιε διαφορέ και αποκλήσει, γιατί κάποιοι φοιτητέ βρίσκουν δουλειά και κάποιοι άλλοι όχι. Νομίζω ότι η ικανότητα να εξεύρει κανεί εργασία εξαρτάται και από τον, ε, το κατά πόσο ένα τομέα ε, έχει ζήτηση και, συγκεκριμένα σε κάθε χώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ένα παράδειγμα στι χώρε της Ανατολική Ευρώπης, κάποιοι τομείς είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί, αλλά όχι σε άλλους τομείς, σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Σε πολύ διαφορετικό βαθμό λοιπόν. Η πληροφορική μοιάζει να είναι σαν ένα σφουγγάρι και απορροφά πολύ κόσμο που έρχεται και από αλλού. Υπάρχουν ε, όμως τομείς που έτσι παραμένουν μάλλον θέσει που παραμένουν κενέ σε άλλου τομεί. Τώρα για τι ευθύνε των πανεπιστημίων προ την κοινωνία ή την κοινότητα εντό τη οποία λειτουργούν. Βεβαίω έχουν ε, ευθύνε τα πανεπιστήμια έναντι τη κοινωνία. Και νομίζω ότι ένας τρόπος να απαντούν έμεσα σε αυτή την υποχρέωση είναι ότι εκπαιδεύουν καθηγητές για την προπανεπιστημιακή εκπαίδευση και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να παράσχουν εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. μέσω των ε, καθηγητών για τα σχολεία, όπως εκπαιδεύονται στα πανεπιστήμια, μπορούν ήδη να κάνουν μια πρώτη κίνηση τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και πολύ σωστά εντοπίσατε ότι ο οικονομικός κόσμος θα πρέπει να συμμετάσχει περισσότερο ακόμα και στον καθορισμό των πανεπιστημιακών προγραμμάτων, των κύκλων σπουδών. Δώσατε ήδη το παράδειγμα των κοινοτήτων στην Φινλανδία που έχουν πραγματικά λόγο και ασκούν επιρροή στο πώς διαμορφώνονται η κύκλη μαθημάτων, τα διδακτικά προγράμματα. Ο κόσμος της οικονομίας, ε, ο οικονομικός κλάδος θα πρέπει να καθορίσει κάποια πρότυπα. Βάσει της αυτονομίας τους λοιπόν τα πανεπιστήμια θα μπορέσουν να καθορίσουν τα προγράμματά τους σεβόμενα ακριβώς αυτά τα ελάχιστα πρότυπα. Βεβαίως δεν είναι απλό να είναι κανείς το ίδιο αποτελεσματικός και στην εκπαίδευση και στην έρευνα και στα θεωρητικά και στα πρακτικά, όμως είναι αξιέπαινη προσπάθεια να επιδιώκει κανεί και τα δύο. Αν μη τι άλλο, σε ένα εισάξιο επίπεδο. Στη Ρουμανία πρόσφατα καθορίστηκε ότι αποφασίστηκε μάλλον ότι είναι το πλέον χρήσιμο το κάθε πανεπιστήμιο αυτόνομα να ορίζει την αποστολή του και την, το περιεχόμενό του και να δρά ανεξάρτητα. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο καθηγητής από τη Βρετανία. Ότι το σκεφτόμαστε λίγο χρησιμοθυρικά το όλο θέμα. Ξέρετε όμως κάτι, πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία. Χρειαζόμαστε φοιτητέ ε, και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ξέρετε, και στο θέμα του κυρίου Σμιτ. Επιχειρήσεις και πανεπιστήμια είναι μια σημαντική πτυχή. Μα ενδιαφέρουν ε, όμω και οι ανθρωπιστικές επιστήμες και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε του φοιτητές να σπουδάζουν αυτές τις επιστήμες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς πάντοτε με τους Αμερικανούς. Σίγουρα έχουν ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν καταπληκτικά πανεπιστήμια, αλλά αυτά τα χρηματοδοτεί η ιδιωτική οικονομία χρηματοδοτούνται από ιδιώτες τα πανεπιστήμια. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την Ευρώπη. Εμείς έχουμε καλά πανεπιστήμια, αλλά δεν έχουμε τα εξαιρετικά πανεπιστήμια που έχουν ίσως στην Αμερική, γιατί υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί. Σε εμά τα πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από τις κυβερνήσεις. Όπως έλεγε ο κύριος Βάτιμο, Πολλές φορές ε, είναι στα πρόθρα της χρεοκοπίας τα πανεπιστήμια. Και δεν θα πρέπει να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Εγώ είμαι από το κρατήδιο του ΣΑΡ και έχουμε ένα γαλλογερμανικό ε, Ινστιτούτο που είναι μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων. Οι φοιτητές ε, σπουδάζουν σε διάφορα πανεπιστήμια και τελικά παίρνουν δύο διπλώματα. Ένα γαλλικό, ένα γερμανικό. Αναγνωρισμένα πτυχία. Βέβαια, φυσικά και πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα. Συνιστώ λοιπόν στους ε, Άγγλους να πάνε σε αυτό το Γαλλογερμανικό Ινστιτούτο αν πάτε στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο πρέπει να μάθετε γαλλικά, αν πάτε στο Γερμανικό πρέπει να μάθετε γερμανικά και έτσι θα μπορέσετε να ενταχθείτε στην ε, Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, εμπειρογνώμονες που ήρθαν ε, στη συνεδρίασή μας για να μας διαφωτίσουν Έχω την αίσθηση ότι άρεσε η ακρόαση αυτή στους συναδέλφους γιατί είπαν ότι έμαθαν πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και για τον εισηγητή μας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ή στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια σύντομη παρέμβαση και μετά θα ακούσουμε και το Συμβούλιο. Η Διευθύντρια του Προγράμματος για τη Διαβίου Μάθηση και τα προγράμματα. Ευχαριστώ Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω την διοργάνωση αυτή τη δημόσια ακρόαση για θέματα που είναι τόσο προσφολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων από τη μια και γενικότερα για τον εξυγχρονισμό τη ε, ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τα πανεπιστήμια και τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν. Γνωρίζουμε ότι η σημερινή κρίση έχει φέρει τα πανεπιστήμια στο επίκεντρο τη προσοχή περισσότερο από ποτέ και έχει δείξει με περισσότερη πίεση και ένταση ότι με τις ταχύτητες των τεχνολογικών εξελίξεων, με τον πολύπλοκο χαρακτήρα της κοινωνίας, των περιβαλλοντικών ε, δυσκολιών όλοι οι παράγοντες απαιτούν από τους ε, φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες ε, και μάλιστα διαβίου. Η ψηλότερη λοιπόν εκπαίδευση σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορέσουμε και να νικήσουμε την κρίση για να ετοιμάσουμε την ανάκαμψη. Ξέρετε ότι το θέμα της ανώτατης εκπαίδευσης θα είναι το κέντρο της ε, ερχόμενης πρότασης της Επιτροπής για την στατικική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα καθορίσει την στατικική μας για την ερχόμενη δεκαετία. Από τη μια, καθώς η εργασία και ο χώρος ε, της απασχόλησης αλλάζουν, ε, χρειάζονται νέες δεξιότητες και προσόντα οι πολίτες. Και βεβαίω έχει επηρεαστεί με την παγκοσμιοποίηση ακόμη και ο κοινωνικό ιστό. Ε, του κόσμου μα. Χρειαζόμαστε λοιπόν δασκάλου, καθηγητέ, ερευνητέ και φοιτητέ που θα είναι άριστοι σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στα καλύτερα ερευνητικά πανεπιστήμια, αλλά το ίδιο και στα περιφερειακά ιδρύματα που επικεντρώνονται στη διδασκαλία και στα προγράμματα που έχουν περισσότερο πρακτικό προσανατολισμό, καθώ και στα τεχνολογικά και επαγγελματικά Ινστιτούτα. Σωστά ε, ανέφερε κάποιο ότι εδώ χρειαζόμαστε ήδη καλύτερη βασική εκπαίδευση για να έχουμε καλύτερη ανώτατη εκπαίδευση. Είμαστε λοιπόν υπέρ της αυξανόμενης διαφοροποίησης των πανεπιστημίων βάσει της ε, ισχύω τους. Δεν νομίζουμε ότι διαφορετικότητα ή η ποικιλία είναι αδυναμία, αλλά μάλλον δύναμη, στοιχείο δύναμης και ευκαιρία. Όλοι οι θυσμοί μοιράζονται κοινέ αξίες και στόχους, αλλά δεν υπάρχει η ίδια αξιολόγηση της έρευνας και της εκπαίδευσης ή το ίδιο μείγμα των ε, ακαδημαϊκών γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων. Θα πρέπει η διοργάνωση των πανεπιστημίων να είναι διαφανής για όλους τους ενδιαφερομένους, ε, κυρίως για τους ίδιους τους φοιτητές, ώστε να μπορούν ε, πληροφορημένοι σωστά να κάνουν μια σωστή επιλογή για τις σπουδές τους. Δεν μιλήσαμε λίγο για την Πολόνια στην ακρόαση αυτή. Αυτό είναι βεβαίω ένα μεγάλο μέρο ε, τη προσπάθειά μα να δημιουργήσουμε και να οικοδομήσουμε την Ευρώπη τη γνώση. Νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία μετά από τόσε μεταρρυθμίσει προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό χώρο ανώτατη εκπαίδευση. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η συνολική εικόνα τη Μπολόνια δείχνει ότι απαιτείται πρόοδο ακόμη και αν η ταχύτητα ή το πεδίο των μεταρρυθμίσεων απικύλουν από χώρα σε χώρα. Και όπω υπογράμμισαν και ο κύριο Κάιζερ και άλλοι ομιλητέ. Νομίζουμε ότι το κέντρο τη προσοχή τώρα θα πρέπει να δοθεί σε συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει εντό των ε, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώ και μεταρρυθμίσει στην ε, χάραξη τη εθνική πολιτική για να αναφέρω μερικέ από τι βασικέ προκλήσει που διαβλέπουμε για το μέλλον. Η μία είναι ότι δεν θα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, πολίτε ε, στην Ευρώπη κατά μέσο όρο που να είναι στην ανώτατη εκπαίδευση, να σπουδάζουν και να είναι και απόφοιτοι, πτυχιούχοι. Ξέρετε ότι στη στρατηγική μα έχουμε θέσει ένα στόχο 40% του μέσου ενήλικου πληθυσμού που να έχει τουλάχιστον επίπεδο ανώτατη εκπαίδευση. Μια άλλη πρόκληση είναι ότι πολλά συστήματα ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη είναι ακόμη κατακαιρματισμένα. Ε, έχουν υπερβολικά πολλού κανόνε και δεν χρηματοδοτούνται αρκετά. Θα πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμαστούν με τις ανάγκες της, εργασίας, της αγοράς εργασίας. Η τρίτη πρόκληση που θέλω να αναφέρω και έχει αναφερθεί επανειλημμένως είναι η πρόσβαση. Μεγαλύτερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, περισσότερη πρόσβαση και εν ώψη ιδίω της γύρανσης του πληθυσμού. Κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε περισσότερους ενηλίκους που θα ήταν καλό να επιστρέψουν στα πανεπιστήμια για να λάβουν περισσότερες γνώσεις ή να ενημερώσουν τις δεξιότητές τους. Η ανάγκη επίσης να αυξηθεί το επίπεδο κινητικότητας για τους φοιτητές ρότα της εκπαίδευσης. Συζητήθηκε και υπάρχουν αρκετά εμπόδια, δυσκολίες. Ξέρετε ότι δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράσινη βίβλο για την άρση των φραγμών της κινητικότητας και ο νέος πρόεδρος της επιτροπή έχει αναφέρει την ευρεία πρωτοβουλία Youth on the Move που σκοπεύουμε να λανσάρουμε για την ενίσχυση της κινητικότητας όχι μόνο στην εκπαιδεύση των φοιτητών αλλά για όλους τους νέους της Ευρώπης. πέραν της διαδικασίας της Μπολόνια και βάσει της ε, προτεραιοτήτων ε, για, τις, ε, για τα πανεπιστήμια της Ευρώπης έχουμε δει τρει ε, τομεί μεταρρύθμιση. Πρώτον, αυτών των κύκλων σπουδών ε, και εδώ το στοιχείο τη αποσχολησιμότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη, το συζητήσαμε ευρέω. Έπειτα η μεταρρύθμιση, η ανανέωση τη ε, διαχείριση των πανεπιστημίων, περισσότερη ανεξαρτησία για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό είναι μέρο τη ατζέντα του εξυγχρονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο τρίτο τομέα σχετίζεται με τη χρηματοδότηση. Με του πόρου. Εδώ χρειάζεται αύξηση και διαφορετικές πηγές πόρων και χρηματοδότησης. Ε, με την, την ατζέντα μα αυτή του εξυγχρονισμού την ε, ενισχύουμε όχι μόνο ενισχύοντα τα κράτη-μέλη στη διαδικασία peer learning, δηλαδή να εντοπίσουν καλές πρακτικέ μεταξύ του και να τι ανταλλάξουν, αλλά και την διαδικασία τη Μπολόνια ενδυναμώνουμε, προσπαθώντας ε, μια διαδικασία που δεν είναι ακριβώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να πετύχουμε του στόχου μα και με το πρόγραμμα διαβίου κατάρτισης, όπου συμπεριλαμβάνεται και το Erasmus και το Erasmus Mundus, το Tempus, τα προγράμματα έρευνας και ασφαλώς τα διευθυντικά ταμεία. Όλα αυτά συντελούν στο σκοπό μας. Σκοπεύουμε να εξακολουθήσουμε αυτή την προσπάθεια εξυγχρονισμού της ανώτατης εκπαίδευσης και θα εγκρίνουμε μια νέα ανακοίνωση το 2011 για τον εξυγχρονισμό της, ανώτερης, της ανώτατης εκπαίδευσης. Πενταετή πενταετούς διάρκειας μετά από αυτήν του 2006 για το ίδιο θέμα. Εδώ λοιπόν ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διαμορφώσουμε αυτό το πολιτικό έγγραφο καθώς να πω και ότι η σημερινή συζήτηση μας έδωσε πολύτιμα στοιχεία για τη μελέτη μας αυτή. Ευχαριστώ. Είναι περίεργο Ευρωπαϊκή Ένωση, Κομισιόν, το Κοινοβούλιο να λένε ότι θα δρομολογήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες ενώ δεν μπορούμε αφού το Συμβούλιο θα μας το απαγορεύσει ή όχι μήπως κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ντάνκεσεν λέει ο κύριος του Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, ως εκπρόσωπος της Ισπανικής Προεδρίας ε, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα κρύψω επίσης ότι είμαι και καθηγητής πανεπιστημίου στη χώρα μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε, που μου την πρόσκληση να συμμετάσχω στην ακρόαση αυτή με τις πολύ διαφωτιστικές παρεμβάσεις που επιβεβαιώνουν πόσο εύστοχο ήταν το εγχείρημα. Στη σύντομη παρέμβασή μου Θέλω να πω ότι ο ρόλος των πανεπιστήμιων είναι πράγματι θεμελιώδης. Στις 25 Ιανουαρίου ο Ισπανός Υπουργός ε, Εκπαίδευσης, ε, παρόν εδώ στην Επιτροπή σας, ε, επέμεινε στο ότι εκπαίδευση είναι ο βασικός πυλώνας στη σχέση μεταξύ των κοινωνιών και ω πονδυλική στήλη για την ανάπτυξη και έλεγε ότι η εκπαίδευση, η επικοινωνία είναι συνώνυμα με την ελευθερία, την ισότητα, τη συνοχή. Σημαντικές αξίε στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Και ολοκλήρωνε λέγοντα ότι η περισσότερη, πιο ποιοτική εκπαίδευση, εκπαίδευση για όλου, θα ήταν άξονα στον οποίο θα επικεντρωνόταν και η Ισπανική Προεδρία. Πράγματι, η Ισπανία ως στόχο της Προεδρίας της έχει θέσει τους εξής στόχους. Πρώτα απ' όλα, η κατάρτιση και η εκπαίδευση πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο του οικονομικού μοντέλου και στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την απασχόληση που είναι υπό εκπτώνηση και ως πόλη αριστείας, έρευνας και επίδειξης θα έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν τα πανεπιστήμια. Δεύτερον, η ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης ε, της εκπαίδευσης και δι της κοινωνικής διάστασης της ανώτερης εκπαίδευσης και της κοινωνικής ευθύνης των πανεπιστημίων. Και τρίτον, η όθηση του ευρωπαϊκού χώρου γνώσης δηλαδή η σύγκληση των δύο σημαντικών χώρων ε, του ευρωπαϊκού χώρου ανώτερης και της εκπαίδευσης και του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας με εξοχρονισμό και εξορθολογισμό των πανεπιστημίων. Αυτοί οι δύο στόχοι νομίζω ότι δίνουν έμφαση στον ειδικό ρόλο των πανεπιστήμιων και γι' αυτό θα επικεντρωθώ και σε αυτούς. Η έρευνα και η καινοτομία σίγουρα είναι οι βασικοί πυλώνε τη νέα κοινωνία τη γνώση. Ωστόσο, η Ισπανική Προεδρία θέλησε να προσθέσει και έναν ακόμη πυλώνα, αυτών τη κοινωνική διάσταση, τη κοινωνική ευθύνη τη εκπαίδευση και συγκεκριμένα ό,τι αφορά τον τομέα της ανώτερης και ανώτερης εκπαίδευσης. Αφετηρία είναι η πεποίθησή μας ότι η προώθηση της κοινωνικής ε, διάστασης, της ισότητα της εκπαίδευσης, ενεργού ηθαγένειας είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες ε, για την κοινωνική ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθούν οι εκπαιδευτικέ αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο να δραματίσει αυτό και στην ε, στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης. Επίσης, ε, πολύ σημαντικά είναι η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη και βιώσιμη οικονομία. Πέραν όμως της κοινωνικής διάστασης υπάρχει και μία ακόμα πτυχή που είναι η κοινωνική ευθύνη. Τα πανεπιστήμια έχουν ως αποστολή τη δημιουργία γνώσεων και την έρευνα, θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να εγγυηθούν και την επιστροφή στην κοινωνία μέσω της καινοτομίας και της μεταφοράς των αποτελεσμάτων. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε την απαραίτητη συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, αλλά και να επιμείνουμε στην αλληλεπίδραση μεταξύ των πανεπιστημίων και του όλου περίγυρου τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος. Παραδείγματο χάρη, δυνατότητε αναπτυξιακή συνεργασία, ε, εθελοντισμού, πανεπιστήμια για του ε, μεγαλύτερου σε ηλικία κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να εμβαθύνουμε προ αυτή την κατεύθυνση και έχουμε προγραμματίσει ένα διεθνέ συνέδριο για το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο Νέα Πρότυπα που θα γίνει στο Σαντιάγο Δε Κομποστέλα 22 και 23 Μαρτίου. από την οπτική γωνία, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να γίνει και μια εσωτερική διαδικασία, η διαδικασία της Μπολόνια δηλαδή, που μας ε, έδωσε τις δυνατότητες που έχει η ανώτερη εκπαίδευση, έθεσε όμως ε, προφανής και τους περιορισμούς που μπορεί να έχει το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν τον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης να τον ενισχύσουμε ακόμη και πέρα από τη διαδικασία της ε, θα πρέπει να τονίσουμε την διδασκαλία, την έρευνα με επίκεντρο τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορών και των επιχειρήσεων. Επίσης, για αυτό το σκοπό θα γίνει ένα φόρουμ συναντήσεων, θα γίνουν επίση πολλέ συναντήσει με πυρογνώμενους πολιτικούς ηθήνοντε, με κοινωνικούς οικονομικού φορεί που συμμετέχουν στο πανεπιστήμιο, συμμετέχουν στην ανώτερη εκπαίδευση. Στόχο θα είναι η αμοιβαία, ε, η αμοιβαία κατανόηση και, καλύτερη γνώση. Θα γίνει επίση και μια συνεδρίαση για τη διεθνοποίηση τη ανώτερης εκπαίδευση στη Μαδρίτη στι 19 και 20 Απριλίου. Υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή της διεθνοποίησης, εξωτερική πτυχή αν θέλετε. Και θα πρέπει να πούμε το εξή. Δεν είναι ε, άγνωστο σε κανέναν ότι ο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερη Εκπαίδευση έχει κινήσει το ενδιαφέρον πολλών περιφερειών του κόσμου και λόγω ε, της τη ε, πολιτική ενισχύσεων με τα προγράμματα επί Εράσμου Μούντου ή το Εράσμου με στόχο την προσέλκυση των μεγαλύτερων ταλέντων. Το πρόγραμμα Tempus επίση που προωθεί προγράμματα εξυγχρονισμού των πανεπιστημίων σε συνεργασία με τρίτε χώρε η Ισπανική Προεδρία θέλει να τονίσει την πανεπιστημιακή συνεργασία και να την προωθήσει πέραν των όριων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε τομείς ε, σε χώρες του πλανήτη με του οποίους έχουμε στενές σχέσεις, η ε, Λατινική Αμερική και Μεσόγειος. Θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε περισσότερο τις σχέσεις μας με τις περιοχές αυτές του κόσμου και θα ενισχυθούν τα όσα γίνονται ήδη, ιδίως στη Μεσόγειο, με αποκορύφωμα την Υπουργική Διάσκεψη Σλοβενία τον Απρίλιο και επίσης μία συνεδρίαση για την ε, Λατινική Αμερική και για τη σχετικά με την ανώτερη εκπαίδευση 27 με 28 Απριλίου στη Μαδρίτη τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών που ζητούν περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη ευημερία. Χωρί εκπαίδευση, χωρί καινοτομία, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι βαθιέ οικονομικέ και κοινωνικέ αλλαγέ. Και ακόμη λιγότερο θα μπορέσουμε να θέσουμε την Ευρώπη σε ηγετική θέση που θα συνάδει θέση αυτή με τις ε, αρχές που τη διέπουν. Πρέπει λοιπόν ε, και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Ε, όντως στο επίκεντρο της Ευρώπης, όπως μας είπε και η πρόεδρος ΠΑΚ, και ως θεματοφύλακες των γνώσεων, ως ναοί της ευφυΐας και της νοημοσύνης, όπως έλεγε ο Μιγγέλ πριν πριν ε, του Πανεπιστημίο της Σαλαμάκα. Με βάση όλες αυτές τις ιδέες λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση των πανεπιστημίων, θα πρέπει να εντείνουμε τα προγράμματα και αυτό θα είναι το επίκεντρο της Ισπανικής ε, Προεδρίας. Η Ισπανική Προεδρία εξετάζει το ενδεχόμενο στο πλαίσιο και του Συμβουλίου του Μαΐου να εγκρίνει δύο έγγραφα τα οποία είναι πάρα πολύ, έχουν πολύ σημαντικές ε, δεσμεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά υποσχόμενα αυτά που ακούσαμε. Πάντως το Συμβούλιο, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για τα πανεπιστήμια, για όλα αυτά τα θέματα και τα ερωτήματα που ακούσαμε σήμερα. Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο Σμιτ, για να κλείσουμε, σας θυμίζω στους συνδεύσεις και τους συνεργάτες προθεσμοί για τροπολογίες έκθεση ΣΜΙΤ 1η Μαρτίου. Κοντά είναι. 1η Μαρτίου. Και όποιος δεν είναι παρόν σήμερα, η βοηθή παρακαλώ να το διαβιβάσετε. Δεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Πρόεδρο. Όταν μου δώσετε την εντολή να συντάξω αυτή την έκθεση, είχα το θάρρος να την αναλάβω, γιατί δεν είμαι ούτε καθηγητής, ούτε επιχειρηματίας, ούτε φοιτητής. Θεώρησα όμως, επειδή είμαι ο μόνος Ολυμπιονίκης στο Κοινοβούλιο, ότι θα έπρεπε να έχω το θάρρος να το αναλάβω. Και μετά διαπίστωσα ότι το θέμα είναι πολύ πολύ πλοκό Και η έκθεση αυτή θα είναι, κατάλαβα, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είχα προβλέψει στην αρχή. Εμπόριο, βιομηχανία, οικονομία, συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Ποια είναι τα εμπόδια στη συνεργασία αυτή. Καθόλου εύκολο το θέμα. Και φυσικά ζήτησα τη συμβουλή και την βοήθεια πολλών άλλων. Σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν σήμερα, εγώ έχω να προσθέσω ότι βρήκα πολύ υλικό για την έκθεσή μου. Παραδείγματος συζητήσαμε με λεπτομέρειες την αυτονομία. Πήρα μια άριστη, ένα άριστο γραπτό κείμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων ακριβώς για το θέμα αυτό. Αυτονομία σε σχέση με τα οικονομικά, την απασχόληση και άλλα. Επίσης, αναφέρθηκε το θέμα ιεράρχησης ή κύρους, σειρά κύρους των πανεπιστημίων και με ποια κριτήρια μπορούμε να κατατάξουμε τα πανεπιστήμια με την ένταση της έρευνας, με τη στενή σχέση που έχουμε με την οικονομία και ακούσαμε και για την κοινωνική ευθύνη τέλος των πανεπιστημίων. Βέβαια η έκθεσή μου δεν αναφέρεται στη χρηματοδότηση, θα το προσθέσω όμως. Τι περιμένουν τα πανεπιστήμια, να έχουν περισσότερους φοιτητές, να ανέβει το επίπεδο της εκπαίδευσης και περικοπή των δαπανών. Δίλημα εδώ. Ακούσαμε για νομικά εμπόδια. Θα τα βάλω και αυτά στην έκθεσή μου για να σας πληροφορήσω και για κάτι άλλο τώρα. Χθες η Επιτροπή υπό την κυρία Πακ ασχολήθηκε με τις κύριες αρμοδιότητες. Οι κύριες αρμοδιότητες για τους φοιτητές αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε τις βασικές αυτές αρμοδιότητες θα πρέπει να τις σκεφτόμαστε συνεχώς. Έχουμε ριζικές αλλαγές, τουλάχιστον τα τελευταία 20-30 χρόνια. Επίσης η πρόεδρος μας είπε να μην συγκρινόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να υπερπαιδίσουμε τα δικά μας εμπόδια. Τι συμβαίνει στο δικό μας χώρο. Τονίζουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ξανά και ξανά και ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ο πιο ανταγωνιστικός πόλος, η περιοχή του κόσμου. Το 2010 είναι το έτος της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Και όταν μια και αναφερόμαστε στις Ηνωμένε Πολιτείε, και εμένα δεν μου αρέσει να συγκρινόμαστε με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πάντως, η στάση του κοινού είναι διαφορετική από αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι το ευκταίο. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, χαριπίν. 40% του εργοτικού δυναμικού υπάλληλοι έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα. Στην Ιαπωνία 50%. Εμείς έχουμε 35%. Είμαστε πίσω. Άλλο παράδειγμα της ΗΠΑ. Ψηλή τεχνολογία. Που απαιτεί τεράστιο δυναμικό καινοτομία και τεχνολογίας. Στην Ευρώπη είναι μόνο 10% πολύ πιο λίγο από το αντίστοιχο ποσοστό της Ιαπωνίας, των μένων πολιτών, ακόμα και της Κορέας. Πολλά τα προβλήματα λοιπόν και πολλά τα θέματα. Η έκθεση που πήρατε θα εμπλουτιστεί με όλα αυτά τα νέα στοιχεία, με τις και με τις τροπολογίες που ελπίζω να καταθέσετε. Και κάτι ακόμη. Αναφέρθηκε και χθες στην Επιτροπή μας. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος μιας επιτροπής όχι επειδή θα έχω την ευκαιρία να δουλέψω με την κυρία Πακ έξι χρόνια συνολικά, αλλά η επιτροπή αυτή εδώ έχει ένα είδος φωτοστέφανο που την κοσμεί. Δεν μπορεί να αποφασίσει ψήφισμα χωρίς να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να δρανίσουμε, να πούμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, σταματάμε. Όχι βέβαια, έχουμε και εμείς ευθύνες. Είμαστε εκλεγμένοι ευρωβουλευτές. Και αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση, κάποια υστέρηση, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στην Κομισιόν και το Συμβούλιο, εμείς πρέπει να πούμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό. Η έκθεσή μου επαναλαμβάνω, σε μεγάλο βαθμό θα εμπλουτιστεί από τις ιδέες και τις σκέψεις και ευχαριστώ όλους για τη σημερινή συμβολή σας και τη συμμετοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Παλ για να μην φοβηθείτε ότι δεν έχουμε κάτι να πούμε, δηλώνω ότι η Επιτροπή μας παίρνει μέρος σε όλα τα προγράμματα στην συναπόφαση. Δυστυχώς ήρθε όταν είχαν αποφασιστεί τα προγράμματα του 2004 η συναπόφαση στην παιδεία, στην κατάρτιση, στα προγράμματα για την νεότητα, πολιτισμό, για τον εθελοντισμό. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ίσως όχι τόσο πολύ όσο ορισμένες άλλες επιτροπές. Αλλά αυτό είναι και η σαγίνη της επιτροπής μας, η γοητεία της. Πολιτισμός είναι κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουν οι άλλες επιτροπές. Είμαστε υποχρεωμένοι να περιοριστούμε κάπως, αλλά όχι στο Λέγιν, όχι στις πρωτοβουλίες μας. Και σε ευχαριστούμε πολύ που ανάλαβες το θέμα αυτό και είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά από τη διαδικασία της Μπολόνια, που δεν ρωτήσαμε κανέναν. Κανένας δεν ρωτήθηκε μάλλον. Υπάρχουν τώρα στοιχεία και για την Κομισιόν και για το Συμβούλιο, ώστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα από ό,τι πήγανε για την Πολόνια, που δεν πήγαν και πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα στη συνεδρίαση. Ξανά, επόμενη συνεδρίαση. Α, συγγνώμη, κάτι ξέχασα. Υπάρχει το σημείο 14. Ευχαριστώ τους ε, προηγούμενους ομιλητές. Συνεχίζουμε με το σημείο 14. Συντονιστές η συνάντησή τους χθες. Σας στείλαμε το πόρισμα με email. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θεωρούνται δεδομένες οι αποφάσεις πέρα της συνέδρια Okay.